αυτά με βάση τις ανάγκες θα πρέπει να ε, παρακολουθούμε πώς θα, γίνεται, πώς, πώς θα χρησιμοποιούνται οι πόροι αυτοί έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, υλοποιήσουμε τους στόχους της χιλιετίας. Η τράπεζά μας ζήτησε από τους μετόχους της να κάνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι να αυξήσουμε το κεφάλαιο, την κεφαλαιογική βάση, στην, ε, στη Σύνοδο Κορυφής ε, του Λονδίνου η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης ε, πήρε αυτή την δυνατότητα και ελπίζω ότι θα γίνει και αυτό στο, θα συνεχιστεί στο Πίτσμπουργκ. Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης πήρε τα χρήματα αυτά. Ελπίζουμε ότι και στο Πίτσμπουργκ θα τα πάρουμε και εμείς. Υπάρχουν όμως, το, αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι ε, υπάρχουν κάποιοι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν το 2010, το 2011. Αυτό είχε αποφασιστεί και θέλουμε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από το 2009. Δηλαδή η υποστήριξη δημοσιονομική για κάποια μεγάλα έργα υποδομής. Πρέπει όμως μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και το 2010-2011. Και ε, γι' αυτό θα πρέπει όλοι να ε, δούμε τι θα κάνουμε και μετά. Ε, διότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο κάναμε είναι να πάρουμε κονδύλια που θα ήταν διαθέσιμα τα επόμενα χρόνια, το 2010-2011, αλλά θα πρέπει και να το χρησιμοποιούμε το 2009. Πρέπει όμως να είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσει αυτή η ροή για να δούμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Πρόεδρος, θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω τον καθηγητή Γκέρ Γουτζ, που έχει κάνει μια πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα έκθεση για μας που θα μα παρουσιάσει την διεθνή απάντηση στην παγκόσμια κρίση και τη μεταρρύθμιση της παγκόσμια χρηματοπιστωτική δομή και παροχής βοήθειας επίπτωση στι αναπτυσσόμενε χώρε. Είναι διε, διευθυντής του προγράμματος ε, Παγκόσμιας Οικονομική ε, Δημοσιονομικής Βοήθειας και Ανάπτυξης στην, ε, στο, στην Οξφόρδη και είναι ειδικό γενικότερα για τα, ιδρύματα του Bretton Woods κτλ. Η κυρία Βούλη. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης έδωσε μια εικόνα του τι παρουσιάζουν τώρα με το όνομα κατεπίγουσα ανάπτυξη του Διεθνές Νοσηματικού Ταμείου Παγκόσμια Τράπεζα ε, και οι διεθνείς οργανισμοί. Δεν είναι όρος αυτός συνηθισμένος ούτε για το Διεθνές Ταμείο, ούτε για την Παγκόσμια Τράπεζα. Κατεπίγουσα ανάπτυξη όμως, τι συμβαίνει ακριβώς. Όπως επεσήμαναν και το Διεθνές Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τραγικές συνθήκες και να σας αναφέρω παραδείγματα. Η δημοσιονομική, η χρηματοπιστωτική κρίση, όπως ξέρετε, ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες την Ευρώπη και πάντως έξω από τον έλεγχο ή την επιρροή ασδήποτε αναπτυσσόμενης χώρας. Πλην όμως, οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης ήταν πολύ πιο έντονες και μακροπρόθεσμες, μακροχρόνιες στις ε, χώρες αυτές. Απότομη αύξηση των τιμών, ε, μείωση ριζική των αποθεμάτων, ε, μείωση ριζική των εξαγωγών ε, ύφεση σημαντική στην ανάπτυξη, μείωση σημαντική των ε, χρηματοπιστωτικών ροών και ριζική περικοπή των εισοδημάτων. Αυτά είναι τα στοιχεία, οι συνθήκε που αντιμετωπίζουν ε, οι πιο φτωχέ χώρε του κόσμου. Αυτή την κατεπίγουσα ανάγκη λοιπόν για την ανάπτυξη την αναγνωρίζουν όλοι οι διεθνεί οργανισμοί και το G20. Θα ήθελα λοιπόν με την ε, παρέμβασή μου να αναφερθώ στην ανταπόκριση του G20 και προχωρώντας την ανάλυση μου να εξηγήσω το τι ακριβώς συμβαίνει τι υποσχέσεις δίνονται και τι συμβαίνει και βέβαια τι επιπτώσεις θα έχουν όλα αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή σας. Η ανταπόκριση λοιπόν του G20 ήταν ταχεία, συντονισμένη και πολλά υποσχόμενη. Υπεσχέθη νέους πόρους για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επιβεβαίωσε ε, υποσχέσεις που είχαν ήδη διατυπωθεί από το G20 για χορήγηση ενισχύσεων, υπεσχέθη νέα κονδύλια για κοινωνική προστασία και για περιορισμό των επιπτώσεων της ε, κρίσης στις πιο μικρές χώρες, 100 δισεκατομμύρια δολάρια νέων κονδυλίων μέσω χρηματοδότησης που θα ερχόταν από τις διεθνείς τράπεζες και έχει ήδη φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ στη δανειοδότηση του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν ακόμη από αυτό το ποσό. Αυτό δείχνει πώς γίνεται η διαχείριση της κρίσης. Κινούνται νέοι πόροι προς τις χώρες αυτές και πάντως περιορίζουν τις επιπτώσεις της κρίσης στις χώρες αυτές. Αλλά ας κοιτάξουμε τώρα και πίσω από αυτή την εικόνα, αυτή την παρατήρηση και ας δώσουμε κάποια στοιχεία πιο ουσιαστικά με ε, παρατηρήσεις από τα κείμενα που έχετε και εσείς λάβει. Η ανταπόκριση του Διεθνούς Ουσματικού Ταμείου λοιπόν σε επίπεδα ρεκόρ όπως είπα δανειοδότησης έχει λιγότερο αυστηρούς στόχους δημοσιονομικούς και πληθωριστικούς, λιγότερες προϋποθέσεις πλέον για τη δανειοδότηση, αλλά από τις ε, συμφωνίες που έχει συνάψει το Διεθνές Νοσματικό Ταμείο ε, ε, στις 18 κατά 22% τα νέα αυτά ποσά πάνε σε χώρες, αυτά τα νέα ποσά του ρεκόρ της δανειοδότησης, πάνε σε ευρωπαϊκές χώρες. 1,6% όπως λένε τα δικά μου έγγραφα, 1,6% της νέας αυτής ε, δέσμης χρηματοδότησης μόνο πηγαίνει σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει τους φόβους που είχε εκδηλώσει με τη δημοσίευματά της Παγκόσμια Τράπεζα ότι θα προκύψουν ε, αναδυόμενες οικονομίες υψηλών εισοδημάτων ε, ύστερα από την κρίση αυτή. Επιβεώνεται επίσης η πρόβλεψη του Εθνικού Μοναδικού Ταμείου που είχε πει ότι μόνο 2% της εξωτερικής χρηματοδότησης, των αναγκών σε εξωτερική χρηματοδότηση των ε, χωρών με χαμηλό εισόδημα θα μπορούσε να εξασφαλίσει. Και με άλλα λόγια, Εάν δούμε την ανταπόκριση του Εθνούς Ομοσπονδιακού Ταμείου, οι υποσχέσεις για νέους πόρους, τα υποτιθέμενα τεράστια ποσά που διατίθενται, δεν έχουν αναλογία στο ποσό το οποίο τελικά φτάνει στις πιο φτωχικές αυτές χώρες, εκείνες που υποφέρουν και πιο πολύ από την κρίση. Ας στραφούμε λοιπόν τώρα προς την Παγκόσμια Τράπεζα. σε σχέση με την οποία το G20 έκανε πολύ μεγάλες, έδωσε πολύ μεγάλες υποσχέσεις ε, για να ρύθμι, μεταρρύθμιση αναθεώρηση του παγκόσμιου συστήματος. Ο Δε Πολ Ζέλικ, ο πρόεδρος της, ε, ο διοικητής της Παγκόσμιας Τράπεζας, είχε ζητήσει από τις χώρες του G20 από τα πακέτα κινήτρων να διαθέσουν το 7% για ένα πακέτο κινητικότητας για την τράπεζα ένα πακέτο μάλλον ευάλω, που θα απευθυνόταν στους ευάλωτους ε, από την Παγκόσμια Τράπεζα. πακέτο όμως το οποίο δεν έλαβε ούτε μία δεκάρα από τις χώρες του G20. Δεν υπάρχουν νέα κονδύλια, μόνο τρία ε, μικρά κονδύλια που θεσπίστηκαν αμέσως μετά την επιστηστική βοήθεια ε, τα μία προσαρμογή θα έλεγα στα οποία έχει συμβάλει, εκ των οποίων στο ένα έχει συμβάλει 43 εκατομμύρια και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των επιπτώσεών της στις αναπτυσσόμενες χώρες και με το ίντα και με το IBRD θα έπρεπε η Παγκόσμια Τράπεζα, δηλαδή με τα δανειοδοτικά της εργαλεία, να κάνει πολύ περισσότερα με βάση τους υφιστάμενους της πόρους. Πράγμα το οποίο θα σήμαινε, και θα ήθελα να σα εξηγήσω, τα εξή δύο πράγματα. Πρώτον, πρώτον η το μεγαλύτερο κομμάτι της ανταπόκρισης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σημαίνει απλώς προκαταβολή υφισταμένων δεσμεύσεων. Δηλαδή μια χώρα έχει ήδη, έχει ήδη ε, διαπραγματευτεί ένα δάνειο για τα επόμενα τρία χρόνια παραδείγματι από την Παγκόσμια Τράπεζα ή το Εθνικό Νομισματικό Ταμείο, προκαταβάλει αυτά τα χρήματα η Παγκόσμια Τράπεζα για, τράπεζα για να διευκολύνει κάπως το κράτο αυτό. Αλλά αυτό οδηγεί ε, σε συνέπεια, στη συνέπεια ότι ε, σε έξι μήνες ή σε ένα χρόνο θα υπάρξει ένα μεγάλο κενό στη χρηματοδότηση και σε χρονική στιγμή μάλιστα όπου η χώρα αυτή θα έχει εγγράψει στον προπολογισμό τη την απορρόφηση κονδύλιων που όμω δεν θα έρχονται. Δηλαδή δημιουργείται λίγο πιο αργά μόνο, με μια μικρή καθυστέρηση μόνο, ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανάπτυξη των κρατών αυτών. Επίση, η Παγκόσμια Τράπεζα θα έπρεπε να ε, ε, απαιτείται, υποτίθεται, να χρησιμοποιεί, να αποδίδει τα εφιστάμενα κονδύλια τη ω συνήθω. Το IDA, λοιπόν, το ε, μέσον που έχει η Παγκόσμια Τράπεζα για να χορηγεί ε, δάνεια στις ε, χώρες χαμηλού εισοδήματος είναι δεσμευμένο κατά τρόπο που ε, του επιτρέπει να διαθέσει κονδύλια μόνο σε χώρες ανάλογα με τις επιδόσεις τους. Δηλαδή τα χρήματα του IDA ήδη έχουν προκατανεμηθεί ε, επί χάρτου τουλάχιστον σε ορισμένες χώρες ανάλογα με τις επιδόσεις τους. Και για μένα και από τις μελέτες που έχω κάνει αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάρουν σχεδόν τίποτα οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τη χρηματοπιστωτική κρίση από το IDA. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός δηλαδή των κρατών αυτών που έχουν ε, πληγεί βαρύτατα από την χρηματοπιστωτική κρίση, είτε δεν έχουν δικαίωμα, είτε δεν ε, έχουν επαρκείς προϋποθέσεις, είτε δεν έχουν επαρκή ανάπτυξη για να λάβουν τα κονδύλια αυτά. Άρα και πάλι και σε επίπεδο Παγκόσμια Τράπεζα παρουσιάζονται σημαντικά κενά στη χρηματοδότηση και πάλι ει βάρο των πιο φτωχών χωρών, των χωρών με το χαμηλότερο εισόδημα. Αυτέ πλήττονται περισσότερο και από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Και βέβαια. Ε, ξέρουμε, λέγεται τέλο πάντων ότι το G20 ανταποκρίθηκε, ανταποκρίθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά. Ναι, αλλά το να αντιμετωπιστούν ε, οι πρώτε ανάγκε που προκύπτουν από την κρίση στην Ευρώπη και τι Ηνωμένε Πολιτείε δεν σημαίνει απαραίτητα ότι στηρίχθηκαν και οι χώρε τη Αφρική, οι πιο φτωχέ χώρε. Αντιθέτω, έχουν λησμονηθεί και απλώ ε, ακούστηκαν κάποια ωραία λόγια χωρί όμω αποτέλεσμα και η πράξη στην ε, ουσιαστική στήριξη των κρατών αυτών. Θα πρέπει να επανέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και να αναλογιστεί και πάλι τι χρειάζεται. Πόρους, ευελιξία και ταχεία ανταπόκριση στην κρίση. Αυτά τα τρία πράγματα χρειάζονται οι χώρες αυτές. Πολύ σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία δέκα χρόνια με την ουσιαστική παρουσία ε, πρωτοκαθεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πιέσεις που άσκησε για τους στόχους της χιλιετίας, της χιλιετίας όπου ήταν ο μεγαλύτερος χορηγός η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο στη χορήγηση ενίσχυσης η Ευρώπη σημείωσε τεράστια πρόοδο προς τους αναπτυξιακούς στόχους αυτούς που τώρα όμως κατακαιρματίζει, αποδιαρθρώνει αυτή η χρηματοπιστωτική κρίση και εδώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Αυτή είναι η κύρια, τα κύρια ευρήματα της έρευνάς μας. Και αν μου επιτρέπετε ακόμη για ένα λεπτό. Η, μεταρρύθμιση του συστήματος διακυβέρνησης επίσης εξετάζεται από την έρευνά μας και τίθεται το ερώτημα εάν αυτό το ζήτημα θα πρέπει κανείς να το συζητήσει και να πιέσει για αλλαγές. Τα τελευταία χρόνια με τη μεταρρύθμιση της, ε, του τρόπου διακυβέρνησης της Παγκόσμιας ε, Τράπεζας και του Διεθνού Προσωματικού Ταμείου ξέρουμε ότι έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις και τώρα βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης αυτά τα διεθνή όργανα χωρίς όμως να έχουν ουσιαστικά μεταρρυθμιστεί. Άρα θα λέγαμε ας τα αφήσουμε για λίγο αργότερα. Θα ήθελα λοιπόν να παρουσιάσω κάποιες παρατηρήσεις και λόγους για τους οποίους θα πέρω επίγοντα χαρακτήρα στην επιτάκυνση των μεταρρυθμίσεων. Οι αναδυόμενε οικονομίε και ιδιαίτερα η Κίνα και η Ινδία, αντιμετωπίζοντα την κρίση, όπω επίση και η Βραζιλία αλλά και άλλε χώρε, έχουν ε, μεγάλη σημασία για την αντιμετώπιση τη κρίση. Η Κίνα είναι χώρα με τεράστια ρευστότητα, τεράστια αποθέματα και αυξανόμενα ενισχυόμενα προγράμματα εμπορίου και αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έτσι λοιπόν το να συμπεριληφθεί και η Κίνα στις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης έχει κρίσιμη σημασία. Ναι. Γιατί όμως η Κίνα είτε σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είτε σε σχέση με την Παγκόσμια Τράπεζα να δεσμευθεί ή να δεσμεύσει ε, πόρους, να δεσμευθεί πλήρως όταν όσο καλές προθέσεις και να έχει την αντιμετωπίζουμε σαν το φτωχό συγγενή ή σαν το κατώτερο μέλος όταν δεν υπάρχει πολυμερής ισοτιμία. G1 ή G7 είναι περισσότερο αυτοί που κινούν τα σκηνιά. Γι' αυτό λοιπόν όταν υπάρχουν ή. Ε, ε, διάφορες ρυθμίσεις δανειοδότησης που οργανώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με βάση τα, το G20 με τεράστιες χρηματοπιστωτικές, με τεράστιες ε, πιστωτικές ε, γραμμές που ε, θα διαθέσουν υποτίθεται κονδύλια, ε, σε αυτές τις πιστωτικές γραμμές δεν υπάρχουν ούτε η Κίνα, ούτε η Ινδία, ούτε η Βραζιλία δεν προβλέπεται ότι θα συμμετάσχουν σε αυτές τις ρυθμίσεις ούτε και θα περίμενε κανεί. Ενώ οι ίδιε αυτέ οι χώρε, η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία, θεωρούν ότι οι χρηματοπιστωτικοί αυτοί οργανισμοί δεν εξυπηρετούν τα δικά του συμφέροντα και μόνο εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μετόχων του G7. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να συμμετάσχουν και να βοηθήσουν στην κρίση αυτή θα ήταν να, το ότι αντιλαμβάνονται πως χρειάζεται για την αντιμετώπιση της κρίσης η δική τους εμπλοκή. Και αυτό θα το πράξουν όταν δουν ότι οι διεθνείς οργανισμοί είναι και δικοί τους οργανισμοί και όχι μόνο του G7. Επίσης, η κρίση αποδεικνύει ότι και οι δύο χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση και ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πιο φτωχών κρατών. Αυτή η μεταρρύθμιση του προγραμματισμού τους έχει διαρκώς παραμεληθεί, αλλά δεν υπάρχει οργάνωση ή οργανισμός στον κόσμο που θεωρητικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών του, εάν δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κύριων πελατών του, των πιο σημαντικών, δηλαδή των πιο φτωχών κρατών των οποίων τα κύρια προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν ταχύτατα. Και επίση η αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και η ανάγκη για αυτού να έχουν στρατηγική διακυβέρνηση, δηλαδή η κύρια δομή τη διακυβέρνηση να παίρνει στρατηγικέ αποφάσει ενώ τα μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα κράτη που έχουν την ιδιοκτησία που ταυτίζονται με την Παγκόσμια Τράπεζα, ε, θα έπρεπε αντί να την κρατούν σε απόσταση και να τις ε, αφήνουν ως περιθώριο μόνο την, ε, τον πολλαπλασιασμό των γραφειοκρατικών δομών, θα έπρεπε να την αφήνουν να αναλαμβάνει τις στρατηγικές αποφάσεις και να δρά κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό, πιο γρήγορο, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις πολιτικές συνέπειες αυτής της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Και γι' αυτό η έρευνά μας προτείνει μια σειρά μέτρων που κατεπηγόντως χρειάζεται να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την χειραφέτηση των οργανισμών αυτών κατά τρόπο ώστε να τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καθηγητά. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε και πολύ κατατοπιστικά. Κύριε Καθηγητά Καπελούκα, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο και πάλι για να απαντήσετε στα όσα είπε η κυρία ε, much. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καθηγητής δεν είμαι ακόμα, αλλά α, ε, ποιος ξέρει. Έχουμε εξαίρετη καθηγήτρια εδώ ενώπιόν μας στο πάνελ. Θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία που ανέφερε η κυρία Γουτς. Το πρώτο είναι το εξή. Η απάντηση των διεθνών χρηματοδοτικών ε, οργανισμών ε, περιορίστηκε από το ίδιο το σύστημα στο οποίο βασίζονται και με το οποίο λειτουργούν. Και δηλαδή δίνουν χρήματα σε χώρες με ένα σύστημα το οποίο ε, βασίζεται στην απόδοση και σε επιδόσεις τους. Καλό είναι αυτό, πολύ καλό <laughs> και πολύ χρήσιμο ε, να δίνεις χρήματα εκεί που ξέρεις ότι θα πιάσουν τόπο και ε, θα δώσουν αποτελέσματα. Αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματικό για να καλύψει τις ανάγκες κάποιων κρατών ε, σε περίοδους κρίσεων. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο που ήθελα να αφήσω. Και το δεύτερο. Η καθηγήτρια κυρία Γουτζ πάνε ιδιαίτερα φιλική και προς εμάς στις περιφερειακές τράπεζες. Ε, είχαμε την ε, ευκαιρία ακριβώ να χρησιμοποιήσουμε εκ των προτέρων πόρους για το 2010-2011, το αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε δύο χρόνια. Δεν μπορούμε ακόμα να το προβλέψουμε. Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι σε μια ε, ήπειρο που στη δική μας πολλές χώρες βγαίνουν από πολέμους. Και δεν είναι ρεαλιστικό να ε, αναμένει κανείς ότι οι επιδόσεις τους θα είναι αρκετά στεναρές για να προσελκύσουν πόρους από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ε, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Γιατί είναι λιγότερο περιοριστικός ο τρόπος δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Βάσει των αναγκών δηλαδή χορηγούν χρήματα. Στην Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης προσπαθήσαμε με τη δική σας υποστήριξη να ε, φτιάξουμε ένα μηχανισμό που είναι μηχανισμός για λεγόμενες εύθραυστες χώρες ε, που είναι γύρω στις 12 και 600 εκατομμύρια περίπου. Αυτό βοηθάει χώρες που βγαίνουν από πολέμους, που δεν έχουν μητρό επιδόσεων αλλά τα παιδιά δεν πάνε ούτε σχολείο ούτε εμβολιάζονται. Είναι όμως πολύ περιορισμένο αυτό το ποσό από τη συνολική πίτα που ε, χορηγούνται τα δάνεια ε, με βάση τις επιδόσεις των κρατών. Ελπίζω και να είναι και αυτό και ένα επιπλέον δίδαγμα από τη σημερινή κρίση. E η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επίσης αναφέρθηκε ε, η ανταπόκρισή της, οπότε για το λόγο αυτό θα ήθελα να καλέσω το λόγο, την, τον εκπρόσωπο γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να του δώσω το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εγώ να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεγάλο βαθμό συμφωνεί με την ανάλυση αντικτύπου της κρίσης που μόλις μας παρουσιάστηκε. Σε αντίθεση με τις αρχικές προβλέψεις που έλεγαν ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν πρόκειται να πληγούν από την κρίση, διότι σχετικά λειτουργούν ανεξάρτητα από τις διεθνείς χρηματαγορές, αλλά τώρα γνωρίζουμε ότι και οι αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται πολύ σκληρά από την κρίση και κυρίως από τις διαδοχικές κρίσεις που ε, έπληξαν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή επισητιστική κρίση, ενεργειακή κρίση, χρηματοπιστωτική κρίση και οικονομική κρίση τώρα. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες για τους διαφόρους διάβλους ε, εκροών ή τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οι κρίσεις φτάνουν στις χώρες αυτές. Ξέρουμε ότι έχουν ε, πληγεί και από τη χρηματοπιστωτική κρίση ως προς τα δάνεια, τα κεφάλαια από τις ε, πιο ε, ενταγμένες αναδύομενες οικονομίες, αλλά και η ενική οικονομική επιβράδυνση έχει εντεκτυπώ και οδήγησε σε μεγάλο περιορισμό της ανάπτυξης και των ρυθμών ανάπτυξης των κρατών αυτών. Έχουν μειωθεί οι τιμές ε, των εμπορευμάτων, το παγκόσμιο εμπόριο και συνεπώς το εισόδημα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, πολύ έντονη ήταν αυτή η ε, κρίση και έχει πλήξει λοιπόν και το εισόδημά τους από το εμπόριο. Αυτές είναι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις, ε, αλλά οι ε, αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν και πολύ σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις και συνέπειες που μπορούν να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους. οι χώρες ε, που δεν έχουν ισοσχελισμένο προπολογισμό δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσει και μεγάλες κοινωνικές δαπάνε. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνο λοιπόν αύξηση τη ανεργία και το Παγκόσμιο Γραφείο εργασία φοβάται ότι ε, θα αυξηθεί η επισφαλής εργασία και ε, θα υπάρχει μεγάλη ανεργία στι χώρες αυτές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι γυναίκε με επιπτώσεις και για τα παιδιά τους. Επιπλέον η κρίση αυτή Όσο μειώνεται το εισόδημα και αυξάνεται η ανεργία, ενέχουν και ένα κίνδυνο πολιτικής αστάθειας, ε, και κοινωνικών ε, ε, ταραχών στις πιο ευάλωτες και εύθραυστες χώρες. Αυτά λοιπόν είναι τα συμπτώματα. Γνωρίζουμε απολύτως ότι ο αντίκτυπος της κρίσεως ποικίλει πάρα πολύ ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια, τις ομάδες πληθυσμού, ανάλογα με το πόσο ευάλωτες είναι και πόσο μπορούν να αντέξουν σε εξωτερικούς οικονομικούς ε, κραδασμούς. Γι' αυτό παρακολουθούμε πολύ στενά τον αντίκτυπο της κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες σε συνεργασία με τις αντιπροσωπείες μας ε, εκεί και πώς απαντούμε Πολύ σύντομα μετά τη Σύνοδο Κορυφή των 20 στο Λονδίνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε μια δέσμη 28 μέτρων στην ανακοίνωση που τυπλοφορείται υποστήριξη των αναπτυσσομένων κρατών για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η ανακοίνωση αυτή λοιπόν εγκρίθηκε και τα περισσότερα από τα μέτρα αυτά ε, τα δέχτηκε και το Συμβούλιο στις 18 Μαΐου ε, στα συμπεράσματά του. Σύντομα να σας αναφέρω διάφορα μέτρα που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κυρίως να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις μας για τη βοήθεια, κυρίως την αναπτυξιακή βοήθεια, ως μοχλό για κινητοποίηση νέων πόρων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ε, δράση ανάλογα με τον κύκλο της οικονομίας και να υποστηρίξει την κοινωνική ανάπτυξη και την απασχόληση, ας πούμε, στη γεωργία, στην πράσινη ανάπτυξη, ε, στο εμπόριο με ενθάρρυνση και κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, συνεργασία για την οικονομική κυβέρνηση, την ασφάλεια, τη σταθεροποίηση και την προστασία των πιο ε, αδυνάτων. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα ποσά, κοινοποιούνται 500 εκατομμύρια από τα αποθεματικά των ε, περιφερειακών προγραμμάτων από το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, με το μηχανισμό ευελιξίας FLEX για την αντιμετώπιση ευάλωτων ε, ομάδων. Αυτά όλα είναι βραχυπρόθεσμα. Είναι ένα εργαλείο που κινητοποιείται γρήγορα και με βάση τη ζήτηση για να βοηθήσουμε, επαναλαμβάνω, τι πιο ευάλωτε χώρες ΑΚΕ που δεν μπορούν να αντισταθούν στεναρά στην κρίση για να διατηρήσουν τις τρέχουσες δαπάνες τους, κυρίως στο κοινωνικό τομέα. Είναι ένα εργαλείο, επαναλαμβάνω, που απαντά στη ζήτηση. Οι εθνικές αρχές των χωρών και υποβάλλουν τα αιτήματά τους και υπάρχουν κριτήρια επιλεξιμότητας. Τα κριτήρια αυτά βασίζονται ε, σε συγκεκριμένους στόχους που είναι τυποποιημένοι και ε, γνωστοί. Για παράδειγμα, υψηλή οικονομική, κοινωνική και πολιτική ε, ευαισθησία, ε, προβλήματα χρηματοδότηση του προπολογισμού. Η υποστήριξή μας μπορεί να βοηθήσει να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά ε, ελλείμματα και επίσης ζητούμε να έχουν και αρκετή δυνατότητα απορρόφησης με ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής βοήθειας και όπου υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας. Ήδη έχει καταρτιστεί κατάλογος κρατών ε, που ε, απευθύνθηκαν στο μηχανισμό αυτό και αυτό τον καιρό έχουμε επαφές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις διάφορες υπηρεσίες για να δούμε ποιες χώρες θα αποφεληθούν από την πρώτη δέσμη μέσα στο 2009 και θα ακολουθήσουν και άλλες το 2010. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και τώρα μπορούμε να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους από την Επιτροπή. Έχουμε κατάλογο αγορητών. Ο κύριο Μίτσελ είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Δόκτωρα Καμπερούκαν και την κυρία Καθηγήτρια για τις παρεμβάσει τους. Θα ήθελα να πω ότι, έχετε, ότι είναι για μένα αποδεκτά σωστά αυτά που λέτε. Δεν έχω αντίρρηση. Απλώ θα ήθελα να πω ότι πρέπει να ξαναβρείτε και την επαφή με την πραγματικότητα, γιατί αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στι ίδιε μα τι χώρε και η δυσκολία που εγώ αντιμετωπίζω ε, τώρα για να σα εξηγήσω είναι ότι έχω Πρόσφατα τύχησε μία τηλεφωνική συνδιάλεξη από το ραδιόφωνο με μία κυρία, σε μια εκπομπή ραδιοφωνική, μια κυρία η οποία αγωνίζεται να σώσει τους καρκινοπαθείς μέσα από μια οργάνωση που έχει κάνει και δεν μπορεί να βρει κονδύλια για να τους σώσει στην χώρα της, στην ίδια στην Ιρλανδία. Και αυτό λοιπόν προφανώς μειώνεται το ενδιαφέρον του κόσμου για την αναπτυξιακή βοήθεια για τις πιο φτωχές χώρες. Και ο κόσμος λέει δεν χρειαζόμαστε μόνο αναδιάρθρωση των δομών και της διακυβέρνησης του Διεθνούς Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά αναδιάρθρωση των δομών και της διακυβέρνησης των ίδιων των χωρών αυτών. Αυτό είναι το πρόβλημα πάνω απ' όλα. Και χρειάζεστε, χρειάζεστε και εσείς οι ίδιοι αυτή την αναδιάρθρωση και την ε, ανανέωση της διακυβέρνησης. Έχουμε τεράστια προβλήματα και ανεργίας και όλα αυτά. Εγώ ήμουν εισηγητής για την ε, κατεπίγουσα επιστηστική βοήθεια πέρυσι και όταν ανακοινώθηκε αυτό το δισεκατομμύριο, το να περάσει σε συμφωνία από το Συμβούλιο ήταν αδιανόητο. Χρειάστηκε να τους πιέσουμε, να τους απειλήσουμε ότι δεν θα εγκρίνουμε τον προπολογισμό αν δεν μεταθέτεταν αυτό το δισεκατομμύριο και πάλι ακόμα και τώρα δεν είμαστε και σίγουροι ότι ήταν επιπλέον ένα δις και όχι ότι αντλήθηκε από κάπου αλλού. Γι' αυτό λοιπόν, ναι βεβαίω και χρειάζεται μεταρρύθμιση και, το, και την προεδρεύουσα από το Συμβούλιο που είδαμε χτε εδώ, την ακούσαμε που μα έλεγε ότι είναι τεράστιο το ζήτημα τη δημοκρατία ω προτεραιότητα προτεραιότητα ε, στο δικό της πρόγραμμα για την ανάπτυξη. Ναι, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αλλά εξίσου σημαντική δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στον αναπτυσσόμενο χώρο, ε, κόσμο. Από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. 1,6% διαβάζω με κατάπληξη, ένα μόνο 6% πηγαίνει στην ε, υποσαχάρια Αφρική. Είναι απαράδεκτο το ποσοστό αυτό. Και από τα όσα άκουσα σήμερα, του πόρου, ε, ευελιξία, ταχύτητα που χρειάζονται, ναι βεβαίω θα ενισχύσουμε όσο μπορούμε ε, του ρυθμού των ε, εξελίξεων. Και για τον δόκτωρα Καμπερούκαν θα ήθελα να ρωτήσω το εξή, γιατί με πολύ μεγάλη έκπληξη είδα στη Ρουάντα ότι η κυβέρνηση τη Ολλανδία και της, του Ηνωμένου Βασιλείου συνεργάζονται στην περιοχή αυτή, μάλιστα με τι τοπικέ κοινωνίε, για να βοηθήσουν ε, στην ανάπτυξη και στην απορρόφηση κεφαλαίων και σε αποτελεσματικές δομές. Εκεί τι κάνετε λοιπόν. Και επίσης θα ήθελα να σημειώσω με ενδιαφέρον την ε, ε, συνεδρίαση του G20 στο Pittsburgh. Ε, ενδιαφέρον διότι είναι 0,20% ή και λιγότερο το ποσοστό που προσφέρουν για τον αναπτυσσόμενο κόσμο οι ΗΠΑ. Γιατί λοιπόν να γίνει εκεί η συνεδρίαση. Δεν είναι η ώρα πια να τους πούμε ότι, ήρθε, ε, ότι πρέπει να τηρήσουν τις, τις υποσχέσεις τους. Όλα αυτά τα ωραία που μας έλεγε ο Ομπάμα πούντα. Πότε θα διαθέσει αυτά που έχει υποσχεθεί για τον αναπτυσσόμενο χώρο. όταν ε, υποτίθεται ότι κάποιος ε, θέλει να σπρώξει προς τα μπρο να βοηθήσει, να προχωρήσουμε, ε, το υλοποιήσει. Και ειδικά στην περίπτωση του Πίτσπουργκ πρέπει η παρουσία και των αντισωμένων κρατών να εξασφαλιστεί. Αυτό για τον δόκτωρα Καμπορούκα. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος ομιλητής ο κύριος Γκάρεντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο μιλητές για την ε, τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή τους. Πρέπει να πω ότι εδώ η κατάσταση είναι παράλογη και για δύο λόγους. Καταρχάς ε, για την θεσμική αντιμετώπιση των αναπτυσσομένων χωρών. Όλοι στην Ευρώπη ας πούμε συμφωνούμε ότι και οι 27 χώρες ε, πρέπει να είναι ενωμένες, ε, δεμένες για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Δεν, ε, μπορούμε, δεν δεχόμαστε ότι κάποιο, κάποια, άλλη χώρα θα είναι, κάποια χώρα θα είναι ξεχωριστή γιατί θα θέσει σε κίνδυνο το όλο σύστημα. Ενώ όμως θεωρούμε ότι το Μπενά ή η Γκάνα μπορούν να γλιτώσουν από μόνες τους Καμία χώρα ΑΚΕ, που είναι και η δική μας η βασική εταίρη στα πλαίσια της ανάπτυξης συνεργασίας, δεν μπορούν να δεν ανήκουν σε καμία από αυτές τις θεσμικές οργανώσεις που αναφέρετε εσείς. Ούτε στις, ε, στο, στους G20, ούτε πουθενά άλλου. Ένα παράλογο αυτό. Δεύτερον, είπατε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνει μόνο, χορηγεί μόνο το 2% για την Αφρική. Η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να πάρει από τα αποθέματα του 2010-2011 για να χρηματοδοτήσει ε, έργα τα οποία τώρα λαμβάνουν χώρα. Λοιπόν, και αυτό παράλογο είναι. Επίσης, μου λένε ότι οι εμπορικές τράπεζες στην Δυτική Αφρική έχουν ε, αντιμετωπίζουν ε, έχουν ε, πλεονάσματα ρευστού και αυτό είναι παράλογο. Από τη μια πλευρά ε, δεν μπορούν να τους δώσουν οι διεθνείς τράπεζες χρήματα. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν επιτόπου χρήματα τα οποία όμως δεν μπορούν να τα πάρουν. Ε, υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε εδώ. Και ένα άλλο σημείο το οποίο είναι παράλογο και αυτό. Ο κατακαιρματισμός των ευθυνών μέσα στα πλαίσια αυτού του που ονομάζουμε ε, διεθνής ή παγκόσμια διακυβέρνηση το Διεθνές Νοσημενωτικό Ταμείο δίνει βραχυπρόθεσμα δάνεια, η Παγκόσμια Τράπεζα δίνει μακροπρόθεσμα δάνεια, η Κίνα συμμετέχει συμβολικά, ούτε καν συμβολικά, ενώ οι δράσεις της οι δράσει της, ε, στην, ε, οι, οι ανεπίσημες βέβαια, στην Αφρική προκαλούν καταστροφές. Όχι διότι ε, παραβιάζει τους κανόνες αντιτάμπινγκ του ΠΟΕ, αλλά γιατί το, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να βάλουν ένα φρένο στην επιδείνωση τη κατάστασης. Εάν τώρα όμως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΠΟΕ μπορούσαν να λειτουργήσουν από κοινού, να συνεργαστούν, αν υπήρχαν γέφυρες συνεργασίες ανάμεσα σε, όλα, αυτά, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε πιο, πολύ πιο γρήγορα, διότι πλατωνικά και μόνο συμμετέχουν ορισμένοι στην, ε, ε, στην όλη συζήτηση. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Τελευταίο, τελευταία παρατήρηση μου λένε ότι για να υλοποιήσουμε τους αναπτυσιακούς στόχους ε, της ε, χιλιετίας ε, πρέπει να έχουμε πάνω από 5% ανάπτυξη στην Αφρική. Ε, ούτως είμαστε κάτω από το 5% και, και αν πέσουμε ακόμα περισσότερο θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα αρνητικής ανάπτυξης. Μπορούμε να ε, κάνουμε όλες τις προσπάθειες του κόσμου. Η Κομισιόν έχει όλες τις καλές, ε, όλη την καλή θέληση να ε, προχωρήσει και να βοηθήσει. Εάν δεν βρούμε μια λύση για τα προβλήματα τα οποία σας ανέφερα, δεν θα έχουμε, κάνει, δεν θα έχουμε καταφέρει τίποτα. Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω, αλλά φοβάμαι ότι θα διαφωνήσω. Εδώ έχουμε τάβρο σε υλοπολείο και εμείς το αρνούμαστε, δεν θέλουμε να το δούμε. Πολύ συχνά πάω στην Ασία, γιατί έχω διάφορες σχέσεις εκεί. Η Κίνα αυξάνεται με ρυθμούς της τάξης του 9%. Η Ινδία αυξάνεται με ρυθμούς της τάξης του 8%. Σήμερα το πρωί το Bloomberg έλεγε ότι η Σιλάνκα, η χώρα που γεννήθηκα, έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη από οποιαδήποτε χώρα σήμερα και είναι ε, ο καλύτερος τόπος για να πάει κανεί να εργαστεί. Αυτά τα λέει ο Bloomberg. Ε, με εξαίρεση την Ινδονησία, όλες οι χώρες της Ασίας αναπτύσσονται με φαινομενικούς ρυθμούς. 75% Ε, της, ανάπτυξης 75% στα επόμενα τέσσερα χρόνια θα έρθουν από την Κίνα. Εντάξει, ο καθένας έχει τη χώρα του και τον ευρωπαϊκό χώρο που συρρυκνώνεται. Εκτός από τη Γερμανία και τη Γαλλία ενδεχομένω, συρρυκνώνεται η Ευρώπη και παρασύρουμε και την Αφρική σε αυτή τη συρρύκνωση. Βασικά δεν έχουμε πρόεδρε μία παγκόσμια οικονομία, δύο οικονομίες έχουμε. Και κάτω από τα ίδια μας τα μάτια, μπροστά στα ίδια μας τα μάτια έχουμε ε, απόκληση ε, και θα πρέπει να σταματήσουμε αυτό το τροπάρι που έχουμε τα 60 τελευταία χρόνια και να μην γελιόμαστε. Όταν μίλησε ο κύριος Μίτσελ για τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι Ιρλανδοί στην εκλογική του περιφέρεια ε, για να ζήσουν οι οικογένειές τους, για να δουλέψουν. Ακούμε τους Ευρωπαίους ηγέτες που λένε πώς θα βοηθήσουν τον αναπτυσσόμενο κόσμο και μετά βλέπουν τα στοιχεία και δεν κάνουν τίποτα. Έχει έρθει η ώρα να απευθυνθούν στους ίδιους τους εκλογείς και να τους ε, καθησυχάσουν, να τους κατευνάσουν. Η ουσία όμως ποια είναι και η αλήθεια. Ο κόσμος ε, που αναδύεται πλέον είναι διπολικός. Εντάξει, είναι για μας μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αλλά θα πρέπει να το δεχθούμε ότι αναδύεται και πάρα πολύ γρήγορα ένας διπολικός κόσμος και θα πρέπει να εμπλακούμε στη διαδικασία αυτή. Αλλιώ, θα ερχόμαστε εδώ στην Επιτροπή μας και θα λέμε ξανά και ξανά όλα τα ίδια και η οικονομία μας να περιορίζεται συνεχώς. Thank you. The floor uh, ο Μπέρμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να διευκρινίσουμε ένα θέμα το οποίο και οι δύο σας αναφέρατε, κύριε Καμπαρούκα και κυρία καθηγητρία. Κύριος Καμπαρούκα, ξεκινώντας, είπε ότι χρειάζεται καινοτομία ως προ τι διαδικασίε. Γιατί συνήθω, ε, όπω είπε ο ίδιο, αν θυμάμαι καλά τα λόγια του, είναι ε, κλειδωμένε μέσα σε δίσκαμπτε διαδικασίε ε, οι χορηγίε, τα κονδύλια. Και εσεί, κύριε καθηγήτρια, επίση είπατε ότι χρειάζεται καινοτομία και μιλήσατε για την ευελιξία, την ταχύτητα και του πόρου που είναι απαραίτητα τρία στοιχεία, τα τρία στοιχεία που πρέπει να εξετάσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν Ενθυμούμε όμως να άκουσα τον όρο Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είτε από, τον ένα, από, από την άλλη ομιλήτρια. Και παρακαλώ να είστε κάπως πιο συγκεκριμένοι ως προς το πώς βλέπετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίζει αυτό το, τους τρεις όρους, δηλαδή ευελιξία, πόρους και κοινοτομία στην ε, διάθεση ή μάλλον την ε, διάθεση ε, κονδυλίων και σε ποιο βαθμό μπορεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεργαστεί με την ε, Παγκόσμια Τράπεζα. Η Πρόεδρος, θέλω και εγώ να μιλήσω. Έχω γράψει δικό μου όνομα στο κατάλογο των Έχουμε ιστορικές ευθύνες νομίζω. Στην παρούσα εποχή. Θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίζω, να υπογραμμίσω το πόσο έχει ξεφύγει από κάθε όριο η δυνατότητα του Bretton Woods και των θεσμών του Bretton Woods να αντιδράσουν στην παρούσα κρίση. 25 δις το χρόνο είχαν στη διάθεσή τους πριν από την κρίση τα ε, κράτη του G7 και η Παγκόσμια Τράπεζα. Ο κύριος Καμπαρούκα είπε ότι για τα αφρικανικά κράτη πριν από το, τη συνεδρίαση του G7 ήταν 5 ή 6 δις διαθέσιμα. Το Διεθνές Νοσηματικό Ταμείο 200 δις είχε πριν από τη συνεδρίαση του G20. Και μετά είπαν ότι θα το ανεβάσω το ποσό αυτό στο 3 Πριν λοιπόν από την συγχώνευση στις 30 Δεκεμβρίου της Merrill με την ε, Bank of America 60 ε, δις διατέθηκαν σε πριμ Αυτά τα χρήματα λοιπόν τα οποία φτάνουν στους φτωχούς είναι πολύ λιγότερα από τους πόρους της Διεθνούς Τράπεζας και της ε, Τράπεζας Αφρικανικής Ανάπτυξης. το πρόγραμμα για να υποστηρίξουμε την, την ευρωπαϊκή οικονομία ήταν ένα δισεκατομμύριο δολάρια και την Αμερική για κάθε μία από τις δύο. Επομένως μιλάμε για χρήματα που είναι, είναι τεράστια ποσά. Και δείτε και τα κέρδη της, ε, Goldman Sachs λίγους μήνες, πριν τώρα πρόσφατα. Δηλαδή μέσα σε λίγους μήνες τα πράγματα επανήλθαν στο, έτσι όπως ήταν στο παρελθόν. Δεν, τα, δεν πήραμε σοβαρά τις αναπτυξιακές προκλήσεις που ε, εμφανίστηκαν. Τώρα όμως έχουμε ακόμα την ευκαιρία κάτι να κάνουμε. Δεν μπορούμε με σταυρωμένα τα, τα χέρια να παρακολουθούμε Ακόμα και με τους ε, λίγους πόρους ε, που έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με τα λίγα χρήματα που μπορεί να δώσει στις ε, χώρες με χαμηλά εισοδήματα. Πρέπει να δράσουμε τους επόμενους μήνες. Ο κύριος Κάσμαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι είναι προνόμιο να σας ακούω και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπατε. Κυρία, κυρία Γούτσο, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεσή σας, η οποία μου έκοψε την όρεξη βέβαια χθες το βράδυ που την διάβασα. Συμφωνώ με όλες τις ε, συστάσεις ε, και νομίζω ότι ε, αυτά τα οποία λέτε ε, ενισχύουν, πρέπει να ενισχύσουν και όλες και να ταρακουνήσουν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πρέπει όλοι να συμμετέχουμε και η Ινδία και η Κίνα ε, η Κομισιό μιλάει για αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων και διακυβέρνηση. Όταν, αλλά πώς μπορεί να μιλήσεις για διακυβέρνηση όταν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μειώνει τις ενισχύσεις. Αυτό είναι παράλογο θα έλεγα. Διακυβέρνηση. Πώς μπορείς να κυβερνήσεις όταν δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις ε, την κατοικία, την, το νερό, την τα υδραυλικά ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, ας ε, επανέλθω σε αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι ε, με τα οποία θα διαφωνήσω και αν είναι εδώ τώρα ο Πρωθυπουργό θα τον συγχαρώ γιατί ε, ενίσχυσε την άυξηση της, της επιδοτής, τη βοήθεια. Λοιπόν, ο κύριος Ντέβα και ένας άλλος συνάδελφος ε, θα πρέπει να ακούσουν ότι ο βιομηχανοϊκός κόσμος ε, δημιούργησε την ε, κρίση αυτή γιατί ήταν αχόρταγος και τώρα αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε από τους φτωχούς να αντιμετωπίσουν την κρίση. Εγώ προέρχομαι από μια φτωχή συνοικία στο Λονδίνο και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μας ε, ε, έπιθε εμάς τους στοχούς να μαζέψουμε χρήματα για να τα στέλνουμε στην Αφρική, στις αναπτυσσόμενες χώρες για να ε, αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Κύριε Μίτσελ, εσεί, με την ιστορία που έχει η Ιρλανδία θα πρέπει να ξέρετε ότι εμεί θα πρέπει να ηγούμεθα τη κοινή γνώμης και όχι να την ακολουθούμε και είχα την ευκαιρία, την, την ευγένεια να σας ακούσω και εσείς θα πρέπει να περιμένετε να με ακούσετε. Κοιτάξτε, δεν έχω ολοκλήρωσα, μπορεί να διαφωνήσετε, αλλά μετά, αφού ολοκληρώσω. Λοιπόν, ο καθένας μας, όλες οι χώρες μας έχουν μια ιστορία. Μια ιστορία όπου ε, αντιμετωπίζουν ε, αντιμετωπίσαμε την φτώχεια ε, και αν δεν μάθουμε από τα παθήματά μας θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Επομένως ας δούμε τι γίνεται στην Αφρική και στην, κυρίως στην περιοχή της νότια, νότια της Σαχάρας. Ε, κάποιοι από εσά μπορεί να μην έχετε διαβάσει ακόμα στην, την έκθεση. και ας δούμε κάποια θέματα, κάποια προβλήματα τα οποία προέρχονται από εμά, από τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, υπάρχουν άτομα που προέρχονται από αυτές τις χώρες ε, και που ε, δουλεύανε στις βιομηχανικές βιομηχανικές χώρες και που έστελναν τα εμβάσματα. Τώρα δεν έχουν δουλειά, δεν στέλνουν εμβάσματα. Και οι κατασκευαστικές εταιρείες εκεί επί τόπου τα, τα, τα, η βιομηχανία έχει κλείσει διότι εμείς δεν αγοράζουμε τα προϊόντα τους και ας δούμε και τις τιμές των, ε, καυσί, των ορυκτών καυσίμων, των ορυκτών, ε, γιατί, ε, που έχουν φτάσει στον ΑΔΙΡ, διότι δεν παράγουμε εμείς, δεν αγοράζουμε. Εγώ θεωρώ ότι ό,τι συμβαίνει σε κάποιους ε, άλλους είναι τόσο σημαντικό σαν, σαν να συνέβαινε σε μένα. Αυτή είναι η ιδεολογία με την, μεγάλη, με την οποία μεγάλωσα και είμαι περήφανος για αυτήν. Λοιπόν, σας, θα σας υποστηρίξουμε και για την μεταρρύθμιση αλλά και για τη συμπληρωματική ενίσχυση και βοήθεια προς αυτές τις χώρες τις οποίες εμείς οδηγήσαμε να φτάσουν στα χάλια τα οποία ε, αντιμετωπίζουν τώρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσίμερ. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε και κύριε Κάσμαν για αυτά που είπατε. Είπατε ε, σίγουρα κάτι ε, με το οποίο συμφωνούμε εδώ πολύ. Θέλω να επανέλθω σε αυτό στην εικόνα που δανείστηκε ο κύριος Δίβα για τον Ταύρο στο Ιωπολείο που δεν μας αφήνει να δούμε την πραγματικότητα. Μα τι μέγεθο έχει πια αυτός ο Ταύρος που πίστεψε κάποτε κανείς ότι οι κρίσει, οι παγκόσμιε και οι σημερινέ και πιο μακροπρόθεσμες μπορούσαν να αποσυνδεθούν ε, από τις επιπτώσει του από τον τρίτο κόσμο. Δεν τα καταλαβαίνω καθόλου αυτά τα πράγματα εγώ. Πώς είναι δυνατόν να διανοούμαστε κάτι τέτοιο και να χάνετε πολύτιμο χρόνο που χάθηκε και μάλιστα ανεπιστρεφτή κατά την άποψή μου για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά, χρήσιμα και εγκαίρως. Ακούω τώρα, λέει ότι συζητούμε για τις ίδιες μας τις χώρες, για τις ε, συνέπειες της κρίσης που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σωστό είναι αυτό και το αισθανόμαστε, αλλά να νομίζει κανείς ότι μπορούμε να το αντιπαραθέσουμε, να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο ε, αντίστοιχο με τις αναψώμενες χώρες και αν θα τις βοηθήσουμε ή όχι, το θεωρώ στραβό αυτό. Στη Γερμανία μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα κινήσαμε δισεκατομμύρια για να σώσουμε τράπεζες που επλήττονται και ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας να αναζωογονήσουμε. Και τώρα καθόμαστε και συζητάμε, και συζητάμε και καιρό για το ένα δισεκατομμύριο για την επιστημιστική βοήθεια και τη διευκόλυνση αυτή. Απίστευτα πράγματα για μένα καμία σχέση δεν έχουν με τα πραγματικά παγκόσμια προβλήματα. Δεν βλέπουμε τις ανάγκες και εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, το καθεστώς μας, την κατάστασή μας, τις χώρες μας και δεν βλέπουμε πώς θα διαλυθεί τελικά ένας κόσμος και δεν θα μπορεί να λειτουργεί. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Πρώτον, επανειλημμένα τονίστηκε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά και τα εμβάσματα ε, προς τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, από τους ε, πολίτες τους που ζουν στο εξωτερικό. Ρωτώ, ποια είναι η στρατηγική τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προσανατολισμός για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Μήπως είναι αντιπαραγωγικό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα εμβάσματα που παγκοσμίω είναι το τριπλάσιο τη αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε συγκεκριμένα και προ την κατεύθυνση αυτή. Και δεύτερη ερώτηση που αφορά και πάλι την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να πούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά την ευθύνη εδώ φέρει ε, το καθεστώς τη ιδιοκτησία για την ανάπτυξη, δηλαδή πώς μπορούμε να δώσουμε πιστώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες με τρόπο που μπορούν να την απορροφήσουν και όχι με τους όρους παγκόσμια αγοράς. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ, κύριο Γκερέρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και τους ε, δύο μιλητές μας και τον κύριο Καπελουκά και την κυρία Γούτση για την παρουσίαση. Ακούσαμε και από τα όσα μας είπαν οι δύο ομιλητές και από τα μέλη της Επιτροπής μας ε, και καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά δύο είναι οι κρίσεις που είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και μάλιστα στενά συνδεδεμένες αλλά δύο είναι οι κρίσεις, πολύ διακριτές σε ε, πολλά στοιχεία. Πρώτον, ως προς την προέλευσή τους, η αιτία της κρίσης για τις αναπτυγμένες χώρες είναι κάποιες συμπεριφορές για τις οποίες ευθύνονται οι ίδιες οι αναπτυγμένες χώρες από τη χρηματοοικονομική απορρίθμιση. Αυτό που κάποτε ο Γκρίσπαν είχε χαρακτηρίσει ε, την ε, ξέφρενη συμπεριφορά των αγορών και με τις διάφορες φούσκες και μεταξύ άλλων ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες στον κατασκευαστικό τομέα. Οι αναπτυγμένες χώρες λοιπόν είναι θύμα ε, μιας κρίσεως που οι ίδιες χώρες αυτές έφτιαξαν και για τις οποίες οφείλονται οι ίδιες. Ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι θύματα μιας κρίσης που δεν προκάλεσαν οι ίδιες. Μειώνονται οι επενδύσεις, μειώνεται η ανάπτυξη, μειώνεται η απασχόληση, μειώνονται τα εμβάσματα και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν, λέω επίσης ότι είναι διαφορετικές οι κρίσεις αυτές και ως προς ε, τις συνέπειές τους. Στις ανεπτυγμένες χώρες αυτές η κρίση ε, είναι τροχοπέδι για την ανάπτυξη για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται να σφίξουν τις ζώνες τους οι κάτοικοι των χωρών αυτών για λίγα χρόνια. Οι συνέπειε όμως για τι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι ότι διακόπτεται η διαδικασία ε, εξόδου από τη φτώχεια. Και η διακοπή αυτή τι θα σημάνει. Ουσιαστικά θα έχουμε μια χαμένη γενιά εκεί μια χαμένη γενιά στην καταπολέμηση της ένδυας, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού. Δύο διαφορετικές κρίσεις επίσης ως προς τις απαντήσεις και την αντιμετώπιση τους. Γιατί υπήρχαν πολλά χρήματα και μεγάλες επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, στην αναπτυγμένη συγγνώμη, ενώ στις αναπτυσσόμενες πολύ λίγοι που επιπλέον είδαν και την αναπτυξιακή βοήθεια ε, των ανεπτυγμένων χωρών να μειώνεται, άρα και το εισόδημά τους. Και επίση είναι διαφορετική η κρίση ω προ τον ορίζοντα εξόδου από την κάθε κρίση. Για ορισμένε ανεπτυγμένε χώρε η κρίση έχει ήδη λήξει. Γαλλία και μερικέ άλλε χώρε, Γερμανία ενδεχομένω, ήδη έχουν καλά αποτελέσματα ω προ το ΑΕΠ τους εξαγγελίες ακούμε ότι στα μέσα του 2010 θα έχει ξεπεραστεί η κρίση. Τελειώνω, τελειώνω. Για τις υπόλοιπες χώρες όμως έχουμε ανεπανόρθωτες σημείες. Και αν κυκλοφορήσει η εντύπωση ότι τελειώνει η κρίση, κινδυνεύουμε να μην αναλάβουμε τη δράση που είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Ένα λεπτάκι μόνο. Χρειαζόμαστε δράση ε, στα οικονομικά ζητήματα, να καταπολεμήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους ε, και μεταρρύθμιση των ε, οργάνων του Bretton Woods. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική συζήτηση και όλοι θέλουν να πούνε κάτι, αλλά μια και δεν έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή μας πρέπει να περιοριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή την παρουσίαση και θα ήθελα να μιλήσω στη γλώσσα μου αν μου επιτρέπετε. Αυτό που μας ε, παρουσιάσατε εδώ και αυτό που είπαν οι συνάδελφοι σχετίζονται με θέματα τα οποία μας απασχολούν εδώ και μήνες. Έχουμε τεράστια απόκληση μεταξύ της πραγματικότητας και των σχεδίων. Πραγματικότητας δηλαδή της υλοποίησης των στόχων της χιλιετίας, το 0,7% του στόχου που δεν καταβάλουν πλέον τα κράτη και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Κάσμαν και με τον κύριο Μίτσελ ότι χρειάζεται αλληλεγγύη και πρέπει και να τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Εγώ μετά τη Βουλγαρία, ε, ε, προέρχομαι από χώρα που μετά τη Βουλγαρία είναι ίσως η πιο φτωχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φρονώ όμως ότι θα πρέπει τις υποσχέσεις μας να τις τηρούμε και αν ε, πρόκειται να συνεχίσουμε να μιλούμε για τις επιπτώσεις της κρίσης Λέγοντα ότι πρέπει να επιβάλλουμε καθεστώ λιτότητα και να περιορίσουμε τις ταπάνες μας. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι για τι αφρικανικέ χώρε, τι πιο φτωχέ χώρε. Περιορισμό των δαπανών σημαίνει απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον λοιμό. Είναι διαφορετικέ οι πραγματικότητε εκεί και τα μεγέθη. Α δώσουμε λοιπόν κάποιε προτεραιότητε με βάση του πόρου που έχουμε στη διάθεσή μα. Βεβαίω και ε, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν είχαν προβλέψει την κρίση αυτή, δεν ήταν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την κρίση αυτή. Αλλά θα πρέπει να εμπλακούμε περισσότερο στη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Έχουμε σε μερικές εβδομάδες τη μεγάλη συνεδρία Διεθνούς Ρωσματικού Ταμείου και Παγκόσμια Τράπεζα και θα πρέπει, πιστεύω, οι ίδιοι αυτοί οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να δώσουν προτάσει και εμεί βέβαια να τι ακούσουμε και να ανταποκριθούμε. Η Αφρική οι χώρε Αφρικής έχουν σημειώσει με μεγάλη πρόοδο, αλλά παραμένουν πολλά προβλήματα. Προβλήματα και κατανομή των κονδυλίων που εισπράττουν. Ο κύριο Μίτσελ μίλησε για το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την επιστημιστική βοήθεια. Αλλά δεν ξέρουμε αν τελικά τα χρήματα αυτά φτάσανε στους γεωργούς για τους οποίους είχαν προβλεφθεί. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει τους στόχους μας να τους διατυπώνουμε με βάση τους πόρους που έχουμε στη θέση μας και να προσδορίσουμε προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε έτσι ο κατάλογος των ομιλητών και θα δώσω το λόγο και πάλι στους προσκεκλημένους για να ακούσω τα δικά του σχόλια. Παρακαλώ. Ο πρόεδρος Καμπαρούκα πρώτα και μετά η κυρία καθηγητή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη του Κοινοβουλίου. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διαθεσή μας θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα όμως να θίξω αυτό που είπε ο κύριος Μίτσελ γιατί είναι σημαντικό. Οι Αφρικανοί που ζουν σε αυτό το παγκόσμιο χωριό ε, έχουν χάσει τα σπίτια τους, ε, ξέρουν ότι έχουν χαθεί σπίτια στην, ε, και θέσει απασχόληση στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και όταν ξεκίνησε αυτή η κρίση, όταν συναντηθήκαμε όλοι αυτοί οι οικονομικοί διαχειριστές στην Τίνιδα, το πρώτο ερώτημα που ετέθη είναι τι μπορούμε να κάνουμε για μας. Για μας. Γιατί βλέπαμε την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα ε, στις διεθνείς προκλήσεις ε, που αναλαμβάνονταν ε, σε διεθνή συνέδρια και το τι γινόταν τελικά. Και είπαμε ότι η Αφρική χρειάζεται οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Όμως οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις ήταν αυτό το οποίο δεν γινόταν στην Ποτσουάνα όλοι συμφωνούν ότι η Μποτσουάνα έκανε όλες τις κινήσεις σωστά. Άρα δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την κρίση η Μποτσουάνα γιατί δεν έκανε τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έπρεπε. Για το ε, πράσινο ακροτήριο επίσης. Ε, δεν μπορούμε να πούμε τα ίδια με την Μποτσουάνα διότι ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί και χάσαν τον τουρισμό και τα εμβάσματα από τους ε, εργαζόμενους στο εξωτερικό. Εάν αυτό συνέβαινε πριν από 15 χρόνια, θα ήταν χειρότερη η κατάσταση. Γιατί τώρα πολλές χώρες έχουν 6-7% ρυθμούς ανάπτυξης λόγω ακριβώς των μεταρρυθμίσεων που έχουν λάβει χώρες στο παρελθόν. Επομένως, συμφωνούμε εμείς οι Αφρικανοί. Αλλά ούτως ή άλλως και οι μεταρρυθμίσεις δεν θα σώσουν την, την Αφρική από τις κλιματολογικές αλλαγές. Ε, οι, οι, οικονομικές μεταρρυθμίσεις δεν θα επιτρέψουν στους Αφρικανούς να πουλήσουν το μαλλί τους, ας πούμε, το μαμβάκι του, συγγνώμη, ε, διότι ακριβώς έχει καταρρεύσει η διεθνής αγορά. Ε, στο Μόντερεϊ, σε μια, σε μια διεθνές συνέδριο, ακούστηκε τι πρέπει να κάνουν ε, οι αναπτυσσόμενες χώρες και για το εμπόριο και για το κλίμα και τα λοιπά. Και τι πρέπει να, τι πρέπει να κάνουν. Και να σας πω ότι χρειάστηκε χρόνος. Αλλά ούτως ή άλλως μέχρι στιγμής στην Αφρική είχαμε προβλήματα α, εσωτερικά. Μετά από 20 χρόνια αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην Αφρική για εξωτερικούς λόγους και δεν μπορούμε να δεχτούμε μία απάντηση που να λέει ότι μόνοι σας οι Αφρικανοί βγάλτε τα πέρα πρέπει να βρεθεί παγκόσμια λύση μία παγκόσμια απάντηση και πρέπει όλοι μαζί να ε, συνεισφέρουμε για τις καινοτομίες. Εγώ θα απαντήσω γι' αυτό, για την καινοτομία και τα υπόλοιπα θα απαντήσει η Γκέρα. Και εδώ είναι μια δέσμευση, αν θέλετε, που έχουμε αναλάβει στην δήλωση της, ε, των Παρισίων για την αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων. Πέρυσι όμως στην Άγκρα που κάναμε μια ανασκόπηση ε, της κατάστασης και να, δούμε, για να δούμε τι έχει γίνει, είδαμε ότι δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ε, επενδύσουμε σωστά αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί πριν από πέντε χρόνια. Και αν γίνουν σωστά, σωστές οι επενδύσεις, νομίζω ότι θα είναι αποτελεσματική η ενίσχυση. Λυπάμαι που δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας λόγω του ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας αλλά αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις μπορεί να μου τις υποβάλλετε διμερώς και θα σας απαντήσω. Για δύο πράγματα όμως εγώ θα ήθελα να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Το ένα αφορά αυτά τα οποία έχουν ήδη ληχθεί και είναι πάρα πολύ, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Μίτσελ στην αρχή της ε, διάσκεψης, της συνάντησης, ε, δηλαδή πώς ε, μπορούμε να αυξήσουμε την βοήθεια σε μακρινές χώρες όταν οι δικές μας ανάγκες δεν είναι ικανοποιημένες. Ναι, ίσως δεν ήταν σωστό Μα εχθέ είπα ότι θα πρέπει να επιβάλλουμε με νομοθεσία το 0,7%. Δεν είναι αυτό το ερώτημά μου. Μιλάτε για χρηστή διαχείριση και σας προσκυρίζω 100% λέει ο κ. Μητσουλαρά. Και εσείς πρέπει να αλλάξετε δική σα τη διακυβέρνηση. Δεν μπορείτε να μπείτε μέσα σε ένα καβούκι και να έχετε μόνο αμυντική στάση για πράγματα μάλιστα τα οποία ούτε καν εγώ ε, δεν ε, είπα και άκουσα το πάθος με το οποίο μίλησε ο κύριος Κάσμαν και τον ακούω και καταλαβαίνω αυτό που λέει, αλλά σε ακούσει και αυτός αυτά που λένε οι άλλοι. Όχι, με συγχωρείτε, ζητώ ε, συγγνώμη ταπεινά για το ότι είπα ότι... Ε, αναφέρθηκα σε κάποιους χρησμούς που δεν είχατε εσείς διατυπώσει, αλλά εν αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα στην Ευρώπη να δράσει κανείς ανεξάρτητα άμεσα και δεν κινδυνεύουν οι δικές σας οι εκλογικές περιφέρειες να καταρρεύσουν από την έλλειψη διακυβέρνηση στην Αφρική. Πλην όμως στην Αφρική έχουν εξασφαλίσει τα τελευταία χρόνια πολύ αργή μεν και πολύ επώδυνη πρόοδο οι χώρες αυτές για καλύτερη διακυβέρνηση. Αυτή όμως η, ε, αυτή όμως η πρόοδος μπορεί να ανατραπεί από τη μια μέρα στην άλλη και να σας εξηγήσω και με σαφή παραδείγματα τι επίδραση μπορεί να έχει αυτό στη δική σας την εκλογική περιφέρεια. Η Σομαλία και η πειρατεία που εκδηλώνεται στη Σομαλία αυτή τη στιγμή οφείλεται στο ότι έχει καταρρεύσει κάθε κρατική δομή μέσα στη Σομαλία και αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα φεύγουν από τη δική σας εκλογική περιφέρεια για να περάσουν στα του Άντεν δεν φτάνουν εκεί που πρέπει. Επίσης, προβλήματα έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα έχουμε ακόμη περισσότερο με την ύφεση λόγω των ναρκωτικών, διότι τα ναρκωτικά περνούν από τη μία χώρα στην άλλη, στον κόσμο, όπου έχουν καταρρεύσει κρατικές δομές με πολύ μεγάλη ευκολία. Εμείς θεωρούμε ότι οι δημοκρατίες μας είναι γερές, αλλά αυτές οι δημοκρατίες στηρίζονται στην λειτουργία την απρόσκοπτη κάποιων άλλων κρατών που τώρα κινδυνεύουν να καταρρεύσουν και αυτό είναι το μήνυμα που έχω να αποστείλω στους ψηφοφόρου σα στην εκλογική σα περιφέρεια. Κάτι ακόμη που θα ήθελα να διευκρινίσω. Για την ανάλυση του ε, ότι το 1,6% πηγαίνει στην υποσαχάρη Αφρική. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι κακοί τεχνοκράτε μα στο Διεθνέ Σωματικό Ταμείο, στου οποίου οφείλεται αυτό το μικρό ποσοστό. Όχι, γιατί αυτό ε, ε, οφείλεται στο γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εκείνη που το ζήτησε από το Ευρωπαϊκό από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε ποιον πηγαίνουν. Να σας δώσω τα στοιχεία από την έκθεση. Η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Ουγγαρία, η Σερβία, η Λευκορωσία, η Λευτονία και η Ισλανδία είναι οι χώρες που ωφελήθηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο μεγαλύτερο ποσοστό. Η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει στα σύνορά τη κατάρρευση, χρηματοπιστωτική κρίση ή γύρω-γύρω από τα σύνορά τη και έχει αποτελέσει πολύ χρήσιμο και ισχυρό εργαλείο το Εθνικό Ταμείο έτσι ώστε να συγκρατήσει τη χρηματοπιστωτική κρίση. Έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και διαδραματίζει το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και γι' αυτό το λόγο οι πόροι του έχουν χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν τι άμεσε συνέπειε τη χρηματοπιστωτική κρίσης σε αυτές τις χώρες. Δεν θέλω κανείς να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση αυτή θεωρώντας ότι τα στοιχεία που σας ε, παρουσιάζω ε, υποδεικνύουν κάποιες κακές προθέσεις σε κάποια χρηματοπιστωτικά όργανα. Όχι. Εσείς ο μεγαλύτερος χρηματοδότης των χρηματοπιστωτικών αυτών οργανισμών και δεν, κάνετε, και δεν κάνουν τίποτα άλλο τα χρηματοπιστωτικά αυτά όργανα παρά μόνο αυτό που εσείς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι μεγάλοι χορηγοί τους ζητούν, θέλουν να πράξουν. Το θέμα όμως είναι εσείς πέραν αυτών των κρατών γύρω και μέσα στην Ευρώπη ε, είστε διατεθειμένοι να στηρίξετε με ενέσει χρηματοδότηση και μικρέ οικονομίε που επίση αποτελούν μέρο τη εντολή του ΔΣΤ Ταμείου που δεν έχει το, χρηματο... το Ταμείο αυτή τη στιγμή ούτε εντολή ούτε πόρου από εσά για να στηρίξετε τι μικρέ αυτέ χώρε. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτή είναι η πρόκληση στην οποία θα πρέπει να δώσετε απάντηση. Για δε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ερώτημα τι είδου ε, ανταπόκριση μπορεί να δείξει. Ναι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να επικεντρωθούμε στα μέσα εκείνα τα οποία μπορούν ταχαίως και αποτελεσματικά να ε, στηρίξουν ε, τις χώρες αυτές στην κρίση. Μιλήστε για 500 εκατομμύρια ευρώ που προστίθηκαν στο Flex και τι ενισχύσει του Flex. Ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτά είναι προκαταβολή υπεσχημένων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να, χρησιμο... να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε πόρου που έχουν ήδη δεσμευθεί και να δούμε όταν εξαντληθούν αυτοί πώ θα καλύψουμε το κενό. Α δούμε επίση ότι αυτά τα χρήματα, αυτέ οι ενισχύσει πάνε σε συγκεκριμένες και στοχευμένες σχεδιασμένες καλά δραστηριότητες όπως την υγεία και την εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε προκαταβάλλοντας ποσά που θα πήγαιναν στην υγεία και την εκπαίδευση μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουμε τα ε, άμεσα, τις άμεσες συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης σημαίνει ταυτόχρονα ότι δημιουργούμε πολύ μεγαλύτερα διαφορετικά προβλήματα στο μέλλον για τις χώρες αυτές. Λυπόμαι που δεν έχουμε άλλο χρόνο και δεν μπορώ να απαντήσω εκτενέστερα στις εξαιρετές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Και τις δυο σας. Και τους δυο σας. Εξαιρετικές παρεμβάσεις σας. Επεξεργαζόμεθα ένα ψήφισμα το οποίο θα απευθύνουμε στη συνεδρία του G20 και προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν τις παρατηρήσεις σας από εδώ και μπρος στις εργασίες μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. με βάση τις, ε, τις πληροφορίες που αντλήσαμε από τη σημερινή συνεδρίαση μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογία. Μόνο προφορική όμως δυνάμει του κανονισμού του άρθρου 156 εκτός και ε, έχει αντίρρηση κάποιο μέρος της Επιτροπής μας. Σας ενημερώνω επίσης ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήρθε σε επαφή μαζί μας για να μας ε, παρακαλέσει να δεχθούμε ε, ομάδα υψηλού επίπεδου εκπροσώπων υπαλλήλων του Διεθνούς Σωματικού Τομείου για ζητήματα χρηματοδότησης των, ε, κρατών, των πιο φτωχών κρατών την προσεχή εβδομάδα. Θα ενημερωθείτε για, το, για τη συνεδρίαση αυτή, για το πού θα λάβει η χώρα κτλ. Αν επιτρέπετε τώρα θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μπορείτε βεβαίως αν θέλετε να μείνετε στη συνεδρίασή μας. Ας κοιτάξουμε τώρα τα θέματα του προϋπολογισμού. We 2010. Έχουμε συντάξει την για τον προπολογισμό του 2010 και πρέπει να προσδορίσουμε προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Θα παρακαλέσω τον κύριο Κέι Μίτσελ να ε, παρουσιάσει το σχέδιό του. Πρόεδρε, μέσα σε συνθήκες αναταραχής λαμβάνω το λόγο. Φαίνεται ότι αν κανείς ε, σηκώσει τη φωνή, τη φωνή για να επισημάνει δύσκολε αλήθειες, όσο αλήθειες και είναι αυτές πάντα ενοχλούν. Έχουμε λοιπόν ένα σχέδιο γνωμοδότηση το οποίο ασχολείται με θέματα χρηματοπιστωτικά και τα, τις μεγαλύτερες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Χρηματοπιστωτική κρίση και συνέπειες των κλιματικών αλλαγών είναι το κύριο μας ε, πρόβλημα και τα δύο άλλωστε υπογράμμισαν ε, η κυρία Γκυνίλα, τα υπεγράμμισε χθε η κυρία Γκυνίλα Κάλσον, η προεδρεύουσα από τη Σουηδία. Μάλλον υπάρχουν πολλαπλέ συνεδριάσεις ε, επιτροπών πρόεδρε αυτή τη στιγμή με στην αίθουσα. μήπω έχω τη δυνατότητα να συνεχίσω ή όχι. Με τη χρηματοπιστωτική κρίση λοιπόν η Επιτροπή πρότεινε να χορηγηθεί ενίσχυση στις χώρες ΑΚΕ χωρίς όμως συγκεκριμένε προτάσεις για τις ε, χώρες DCI ενώ οι περισσότερες χώρες, οι περισσότεροι άνθρωποι που πλήξαν οι πιο φτωχοί άνθρωποι ζουν στην Ασία. Ίσως λοιπόν θα πρέπει μέσα στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των ε, ε, κειμένων στρατηγικής για τις χώρες της CIA να συμπεριληφθεί αυτή η πρόταση. Και εγώ ετοιμάζω σχετικά έκθεση για την Επιτροπή. Αλλά αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε από τον έναν για να δώσουμε στον άλλον. Το DCI ήδη προβλεπόταν να ενισχυθεί για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των πολιτών της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής πριν καν να ακουστεί η λέξη χρηματοπιστωτική κρίση ή οικονομική κρίση. Οι ανάγκες που προκύπτουν από την κρίση είναι επιπρόσθετες και για να αντιμετωπιστούν πρέπει να προσθεθούν νέα κονδύλια. Χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση. Η νέα κρίση και γι' αυτό απευθύνομαι προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρωτήσω πώς θα βοηθηθούν οι χώρες αυτές ώστε να αντιμετωπίσουν την κρίση. Δεύτερο ζήτημα, Πρόεδρε, οι κλιματικές αλλαγέ, όπου οι πόροι που βλέπονται από τον προπολογισμό δεν αρκούν για να αντιμετωπιστούν τεράστιες ανάγκε προσαρμογής και περιορισμού των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών. Εγώ προτείνω επιπλέον ποσά 55 εκατομμυρίων ευρώ ε, βάσει και των πληροφοριών που λάβαμε χθε το βράδυ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα καταθέσω σχετικά προφορική τροπολογία. Έστω και αν γνωρίζουμε ότι πολύ, ε, πολύ περισσότερα κονδύλια θα χρειαστούν πριν, την ολοκλήρωση, πριν το κλείσιμο των δημοσιονομικών προοπτικών του 2013, όπου και πάλι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει ηγετικό ρόλο για να εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους. Ξέρω βεβαίω ότι δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια. Αυτό όμως ε, οφείλεται στο ότι οι δημοσιονομικές ε, προοπτικές επιβάλλουν πολύ χαμηλά όρια για τις δαπάνες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τίτλο 4. Το σχέδιο γνωμοδότησης επαναλαμβάνει την έκκλησή μας για ανατροπή, για αναθεώρηση καλύτερα αυτής της συμφωνίας. Και εν τέλει θα ήθελα ιδιαίτερα να ε, διαμαρτυρηθώ για την πρακτική που ακολουθήθηκε και φέτος, αλλά όπως και πέρσι, τη ε, διάθεση δηλαδή στην ε, κίνηση της δημοσιονομική διαδικασία ασφαλμένων πληροφοριών που ε, μας, ανάγκασε να περιμένουμε ε, και να καθυστερούμε τη δουλειά μας μέχρι ότου διατεθούν πλήρες πληροφορίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στα θέματα του προπολογισμού εχθές ε, στη συνεδρία του Κοινοβούλου και έλαβα email εχθές το βράδυ για να συμπληρώσω την εκθεσή μου. Δηλαδή λιγότερο από 24 ώρες πριν από την προβλεφτή σε ώρα για την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας. Δεν είναι δυνατόν τελευταία στιγμή να μου έρχονται συμπληρωματικές πληροφορίες και έχω βεβαίω διαμαρτυρηθεί ήδη. Για άλλη μια φορά δεν επαναλαμβάνω την ε, διαμαρτυρία μου και μέσα στη συνεδρίαση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με νομοθετική, αρμοδιότητα σε επιτροπή, όχι με κάποιο όργανο ε, συζητήσεων μόνο. Και πρέπει να μας ε, υπολογίζει με σοβαρότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μας διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορούμε να παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και εγώ κύριε Μίνσελ, ο κύριο Στίβα. Παρακαλώ τους συναδέλφους να λάβουν το λόγο για τη συζήτηση. Τέις Μπέρμαν, πολύ σύντομα πρόεδρε. Ο συνάδελφος Μίτσελ νομίζω έχει κάνει καλή έκθεση. Η δική μας δουλειά είναι ως Επιτροπή Ανάπτυξης να επαναφέρουμε το ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στα λογικά πλαίσια και στα δίκαια πλαίσια. Καλά το έχει κάνει ο εισηγητής. Η συνάδελφος Ζαμπόσκα έχει κάνει κάποιες ε, τροπολογίες και με κρυφό τρόπο και ύπουλο θεεί τα δικαιώματα στα αναπαραγωγικά ε, υγεία των γυναικών ε, και θεεί για τις εκτρώσεις, για τις αμβλώσεις. Αυτές είναι τελείως απαράδεκτες τροπολογίες και δεν μπορούμε να τις δεχτούμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ζεπόσκα, ε, ε, θα ήθελα να δικαιολογήσω τις τροπολογίες μου. Στις ε, συνεισφορές μου, σε όλες τις εκθέσεις μου, ανέκαθεν υποστήριζα την υγεία των γεγονών, την υγεία των μητέρων, αλλά δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθεί τις, αυτές τις πρακτικές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρακτικές όπως οι αμβλώσεις, παραδείγματος χάρη. διότι αυτό δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς και υπέβαλα τις τροπολογίες αυτές. Διότι υποστηρίζοντας τις αμβλώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, επεμβαίνουμε στις αρμοδιότητες των κρατών αυτών. Κύριος Μίτσελ, δεν ξέρω αν δεν το κατάλαβα καλά. Οι τροπολογίες αυτές μιλάνε για ε, ε, αναγκαστική άμβλωση. Ποιο είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω. Η κυρία Σαμπόσκα κατέστησε σαφές ότι η διατύπωση η διατύπωση των τροπολογιών της είναι υπέρ των ε, μάλλον τις αναγκαστικές αμβλώσεις ε, δεν μπορεί να τις ε, καταδικάσει κανείς αλλά το πρόβλημα είναι για τις υπόλοιπες τι γίνεται καταδικάζουμε τις άλλες αμβλώσεις κύριος Μίτσελ δεν έχει σημασία ποια είναι η θέση της κυρίας Αμπόσκα ή οποιοδήποτε άλλο το πρόβλημα είναι τι θα λέει η νομοθεσία εδώ μιλάμε για αναγκαστικές αμβλώσεις δεν ξέρω τι γίνεται, πώς, ποια είναι η, η ερμηνεία που έδωσε στο κείμενο, αλλά εγώ μιλάω για αναγκαστικές αμβλώσεις και το έχουμε υποστηρίξει και στο παρελθόν. Κύριο Ντέβα, μιλάμε, κύριο Ντέβα, μιλάμε για τις τροπολογίες που έχουμε μπροστά μας. Και νομίζω ότι υπάρχει και, ένα, και μια προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών για αυτή την έκθεση. Το πρόβλημα είναι να δούμε. Πρέπει να δούμε τι λέμε, τι, θέλουμε. Η φωνή του Βατικανού ακούστηκε με σαφήνεια σήμερα. Η κυρία εκεί στο βάθος. Έχω το λόγο. Α, Πολύ γρήγορα έγινε αυτό. Εγώ απλώ ήθελα να μπω στον κατάλογο. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για την, για την άμβλωση, άρα θα περιμένω να, έρθει, να, να λύσουμε το θέμα των αμβλώσεων και μετά. Κύριος Κούσμαν, ευχαριστώ. Δεν θα, δεν θα αναφερθώ ούτε στον Πάπα ούτε στο Βατικανό, αλλά θα πω το εξή. Πρέπει να δούμε την τροπολογία που έχουμε μπροστά μα. Αλλά πρέπει να δούμε και τι συνέπειε όμω. Ποιε είναι οι συνέπειε οποιασδήποτε τροπολογίε και νομίζω ότι η κυρία Σαμπόσκα ε, υπογράμμισε αυτές τις συνέπειες. Ε, η πρόθεση ε, της πολιτικής μας ομάδας και άλλων ομάδων είναι να καταψηφίσουμε τις τροπολογίες. Εάν κάποιος ε, ε, μας πείσει ότι προστατεύουμε τα δικαιώματα των γυναικών να διαλέξουν, μπορεί να αλλάξουμε. Αλλά υπό το φως των δηλώσεων της κυρίας Αμπόσκα που προβάλλει το μέλλον, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτή την τροπολογία που αφαιρεί στο κάτω-κάτω το δικαίωμα από κάποιο άτομο να επιλέξει. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μου συμμερίζεται απολύτω στι επιφυλάξει που εξέφρασε τώρα η σοσιαλιστική ομάδα. Διαβάζοντα δηλαδή και εγώ αυτέ τι τροπολογίε, αισθάνθηκα αποτροπιασμό στο θέμα αυτό. Συμφωνούμε απολύτω με το όσα είπατε κι εσεί. Αν μου επιτρέπετε πολύ σύντομα, Πρόεδρε, για να απαντήσω. Θεωρώ ότι όσοι στην έκθεση ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να απαγορευθούν, ότι εκείνοι που είχε ζητήσει να απαγορευθούν από, την έκθεση αυτή οι ε, καταναγκαστικές αμβλώσεις ήταν η κυρία Γκόμες ε, στην προηγούμενη θητεία και δεν νομίζω ότι ήταν της άκρας δεξιάς οι θέσεις της. Ο Πρόεδρος, κοιτάξτε, ψηφίζουμε με βάση αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Λάθος σας είπα ότι έχουμε την ψηφοφορία το Σεπτέμβριο. Τώρα ψηφίζουμε, σήμερα λοιπόν. Σε 10-15 λεπτά θα ψηφίσουμε και ψηφίζουμε με βάση το κείμενο που έχουμε μπροστά στα μάτια μας, όχι με αυτό το οποίο θεωρούμε ότι ενδεχομένω είναι η πρόθεση κάποιου. Ο κύριος Κάσμαν. Κύριε Ντέβα, επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω κάτι που είναι προφανές, ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τις σκεμμένες σημεί επιπτώσεις αποφάσεων και επιλογών της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου ο κύριο Μίτσελ. Πρόεδρε, βαρέθηκα να ακούω αυτέ τι ανοησίε. Η κυρία Γκόμε πέρσι κατέθεσε την τροπολογία αυτή. Η κυρία Γκόμε ήταν εκείνη η οποία κατέθεσε την τροπολογία αυτή και ομόφωνα, αν δεν με την είχε υποστηρίξει η Επιτροπή μα. Το πρόβλημα είναι ότι η κυρία Ζαμπόρσκα, καταθέτοντα την ίδια τροπολογία, προκαλεί αντιδράσει από ορισμένου που θεωρούν, κάνουν προβολέ ε, ότι και έτσι υποστηρίζουν τι καταναγκαστικέ αμβλώσει και όχι τα δικαιώματα των γυναικών σε επιλογή. Μόνο την καταναγκαστική άμβλωση υποστηρίζουμε τη συμπεριφορά του αυτοί οι άνθρωποι. Η κυρία Γκόμε ακριβώ την ίδια διατύπωση είχε, είχε περιλάβει στην τροπολογία τη ε, πέρυσι. Ακριβώ την ίδια διατύπωση. Παρακαλώ κύριε Μπον. Εντάξει, μια που όλοι αρχίσαμε να ερμηνεύουμε τα λόγια ενός του, όλου, του άλλου, α εξηγήσω και εγώ ξεκάθαρα ότι οι σοσιαλιστές δεν θα υποστηρίξουν τις καταναγκαστικές αμβλώσεις ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι, λέει ο κύριο Δίβα. Οι σοσιαλιστέ λοιπόν δεν υποστηρίζουν τις καταναγκαστικές αμβλώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε. Χωρίς μικρόφωνο. Έχω να διατυπώσω μια πολύ αυστηρή κατηγορία κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαθε... Να σημειώσω μάλλον μια πολύ αυστηρή κατηγορία που διατυπώθηκε κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν επιτρέπει ε, με τι πληροφορίε που διαθέτει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρκετό χρόνο για μελέτη των υποθέσεων και το λήψη αποφάσεων. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μάρτιν Πέντιγκτον, επικεφαλή του τμήματο ε, για την διαχείριση και την εφαρμογή σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση των εξωτερικών προγραμμάτων ενίσχυση αλλά και των ε, ενισχύσεων στο χώρο των προενταξιακό που γίνεται, γίνονται, διατίθενται χάρη στι αντιπροσωπείε μα και τι αποστολέ μα στι εν λόγω χώρε. Α ανταποκριθώ λοιπόν πρώτα στι παρατηρήσει του κυρίου Μίτσελ ω προ τι πληροφορίε που του δώσαμε. Όπως στο email που του έστειλε αυτά το βράδυ, του επεσήμανα άλλωστε, ε, πρέπει να ετοιμάζουμε πολύ νωρί το προσχέδιο του προπολογισμού. Υποβάλλεται μεν στο κοινοβούλιο το Μάιο, πλην όμω έχουμε ξεκινήσει τον Ιανουάριο εμεί την προπαρασκευαστική εργασία. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο οι πληροφορίε στο προσχέδιο του προπολογισμού ίσω να μην είναι τόσο φρέσκε ή τόσο ενημερωμένε. Από την άλλη βέβαια πρέπει να είμαστε και σύντομοι στι πληροφορίε που διαθέτουμε. Ασφαλώς αντιλαμβάνομαι ότι τον αποστολή ε, διορθωτική επιστολή την παραμονή, επειδή ακριβώ αυτό το πράγμα όμω ε, απεφασίστη εχθέ σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ το ταχύτερο δυνατό το απέστειλα στον κύριο Μίτσελ. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι οδηγεί σε δυσκολίε και ορισμένα ζητήματα τα οποία συζητούνται στην Επιτροπή. Όμω, είναι θέματα που συστήσαμε και εχθέ ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, ομολογώ και εγώ ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τον ε, συντάκτη να ε, μελετήσει και να ανταποκριθεί 100% στις, στα νέα αυτά στοιχεία. Ζητώ συγγνώμη για την εξέλιξη αυτή, για τα συμβάντα αυτά. Βεβαιώ τόσο τον, το συντάκτη όσο και την Επιτροπή ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να έχουμε την βέλτιστη δυνατή συνεργασία και να σας συνεπικορούμε στο έργο μας, το έργο σας. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι με πολύ μεγάλη χαρά θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά ε, και λεπτομερέστερα κατηδία με τον κύριο Μίτσελ αν το ε, επιθυμεί για να ε, διασκεδαστεί οποιαδήποτε δυσθυμία. Επίσης, πολύ σύντομα, κάποιες σύντομες αναφορές που ακούστηκαν σήμερα το πρωί για το πρόγραμμα επιστημικής βοήθειας που συμφωνήθηκε πέρυσι και την αδυναμία εξέβρεσης πόρων θα θυμάστε ίσως ότι ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε για πρώτη φορά την πρόταση για το μέσο επιστηστικής βοήθειας. Ελπίζαμε ότι θα γινόταν η χρηματοδότηση, ότι θα εξασφαλιζόταν η χρηματοδότηση από τον τίτλο 2, δηλαδή κονδύλια τα οποία δεν ήταν απαραίτητα για την ενίσχυση των Ευρωπαίων αγροτών θα μπορούσαν να απευθυνθούν στους αγρότες των φτωχών κρατών του κόσμου. Δεν έγινε δεκτή όμως η πρόταση αυτή και γι' αυτό κάναμε ό,τι περούσε από το χέρι μας για να εξάγουμε τα κονδύλια από τον τίτλο υπαριθμών 4, κάθε μέσον με τήλθαμε, όπω είπα, συμπεριλαμβανομένη και τη οργανική συμφωνία. Η ε, διάθεση αυτών των κονδυλίων προχωράει πολύ καλά. Πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ έχουμε ήδη κατά νήμη. Έχουμε ήδη δεσμεύσει πάνω από 700 και ελπίσουμε να φτάσουμε στα 850 σε δεσμεύσεις μέχρι το τέλος του έτους. Και θα ε, αξιοποιήσουμε όλες τις πιστώσεις πληρωμών, τα 450 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε στη διάθεσή μας. Ξέρω ότι ο κύριος Μίτσελ επιθυμεί να, ε, θα επιθυμούσε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να δείξει ότι ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια διεθνή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Και ομολογώ και εγώ ότι ναι, μπορούμε να το πράξουμε αυτό, αλλά όσο προχωρούμε τόσο πολλαπλασιάζονται και τα προβλήματα και γι' αυτό προσπαθούμε να δείξουμε ότι βοηθούμε και τις χώρες που καλέπτονται από το μέσον DCI στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, χώρες οι οποίες ήδη έχουν εισπράξει ενίσχυση από το μέσο επιστημικής βοήθειας που όμως επειδή ακριβώς η κρίση είναι τόσο περίπλοκη και πολυδιάστατη δεν μπορούμε να τις αποκλείσουμε από το DCI και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συνοδευτική και τροποποιητική επιστολή την οποία ετοιμάσαμε όλοι σήμερα καταγράφει την κατάσταση στον τίτλο 4 αναφέροντας ταυτόχρονα και τους τρόπους που ενδεχομένως να μετέλθουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη διαθέσιμων πόρων. Αλλά δεν είμαστε και ε, ε ταχυδακτηλουργοί να βγάζουμε λαγούς από τα καπέλα μας και ως εκ τούτου θα πρέπει να βρούμε κάποιους πρακτικούς και ρεαλιστικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Θα κάνουμε στη μεσοπρόθεσμη, ε, έρευνα, ε, μεσοπρόθεσμη ανάλυση, επισκόπηση των κρατών και των κονδυλίων που έχουμε στη θέση μας για να μπορέσουμε ίσως να καταλήγουμε διαφορετικά τις ε, πιστώσεις που διατίθενται. Επίσης η αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση τα τελευταία χρόνια είναι ένα ζήτημα το οποίο μας δεσμεύει ε, ό,τι έχουμε δηλαδή εισπράξει το απορροφούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Άλλωστε και οι Προεδρεύουσα χτε ε, το επισήμανε. Και μπορούμε να σας δώσουμε λεπτομερείς ε, πληροφορίες με το εγχειρίδιο Better Fast and More, καλύτερα, πιο γρήγορα και περισσότερα, που θα σας αποστείλουμε πολύ γρήγορα. Για το Ταμείο το σχετικό με την ε, Παλαιστίνη και τις κλιματικές αλλαγές που προβλέπονται με ένα προσυπόμνηση για τις ε, προβλεπόμενες συστήσεις με τον ΠΟΕ για την μπανάνα. Είναι άλλα σημεία που θα ήθελα να σας αναφέρω. Έχω και άλλες προτάσεις για το σχέδιο ψηφίσματος. Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να θεωρείτε και εσείς ότι έχω καλύψει τα κύρια ζητήματα ζητήματα, αλλά ασφαλώ θα χρειαστούν ίσω πιο λεπτομερεί απαντήσει και σχόλια. Για τον προπολογισμό και τις τροπολογίε σχετικές με τον προπολογισμό. Θεωρούμε ευπρόσδεκτες και ευχαριστούμε την αποκατάσταση, για την αποκατάσταση των προτάσεων ε, του προσχεδίου σε περισσότερους ε, τομείς. Για τα θύματα βιασμών θα θυμάστε βέβαια και την ακρόαση του κυρίου Ντεγκούχτ ε, την Τρίτη που επίσης κατέγραψε το θέμα αυτό ως προτεραιότητα. Επίσης αναφέρομαι και στις αξιολογήσεις που μάλλον καλύπτονται από τον DCI. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις αξιολόγησης από πλευράς μας των σχεδίων. Θα δείτε τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων στην αίτηση έκθεση μας που έχει ήδη δημοσιευθεί. Στο 55-29 για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα θέλαμε περισσότερες διευκρινήσεις γιατί πρόκειται για ένα σημείο το οποίο μας έχει γεννήσει δυσκολίες σχέση με άλλες διεθνείς δραστηριότητες, ιδιαίτερα το UNFPA και το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Μέσο ε, για τη Σταθερότητα και τη Δημοκρατία. Υπάρχουν διαφορετικές ε, και εξειδικευμένες διατάξεις. Για την τροπολογία 5502 υπάρχει ήδη πρόβλεψη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για τέτοιες δράσεις. Για δε την 5532 ε, περιμένουμε να αναλυφθεί όχι πρωτική δράση, αλλά να χρηματοδοτηθεί δράση από το ICI+. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Όπως είπα, θα συνεργαστούμε στενά και με τον κύριο Μίτσελ από εδώ και μπρο, έτσι ώστε να τον βοηθήσουμε στην ε, επιτέλεση του έργου του, στον βαθμό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτές τις τόσο ε, ενδιαφέρουσες και... Ε, Ελπίζω ότι το, η Κομισιόν δεν θα πιέσει άλλη φορά το Κοινοβούλιο να δεχτεί κείμενα χωρίς ε, να ε, έχει κάποια χρόνο στη διαθεσή του για να αποφασίσει. Uh, chair, my Κοιτάξτε, ήμουνα στον κατάλογο για, την, για τον προϋπολογισμό και το κλείνουμε το θέμα αυτό. Μετά την αλλαγή της Προεδρίας. Να κάνει ένα πρόβλημα. Μπορεί να πάρετε το λόγο τώρα. Κοιτάξτε, για να απαντήσω στην τελευταία παρατήρηση που έκανε η Κομισιόν, για το 5502 για την τροπολογία στη Συμφωνία της Κοπενχάγης για την αλλαγή του κλίματος των πρασίνων θα ήθελα να υποβάλω μια προφορική τροπολογία που και κάνουμε την πρόταση αυτή την κάνουμε ε, πιλωτική πρόταση γιατί υπάρχουν κάποιες τεχνικές ελλείψεις γιατί πιστεύουμε ότι με την τροπολογία αυτή μπορούμε εμείς οι πράσινοι να δείξουμε στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο ότι θέλουμε μια πραγματική χρηματοδότηση για την αλλαγή του κλίματος σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και ε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο εισηγητής υποστηρίζει την πρότασή μου. Και τώρα θα σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των συντονιστών της 3ης 1ης Σεπτεμβρίου προς έγκριση από την Επιτροπή μας. The Ορισμός ε, εισηγητών. Το ΕΛΚ να έχει δύο συντονιστές, τον κύριο Κάσμαρε και τον κύριο Μίτσελ. Ναι, εκπροσωπούν για όλα τα θέματα ε, το ΕΛΚ. Δύο συντονιστές. Επίσης, δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας επιπλέον, Ελάφρυση της στόχιας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, ο δρόμος προς τα εμπρός και ανατέθηκε στο ΕΛΚ για δύο πόντους αυτή η έκθεση. Δεύτερη αναθεώρηση της εταιρικής σχέσης ε, ε, και Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοτομού η πρόεδρος θα κάνει την έκθεση αυτή χωρίς κανένα πόντο. Γνωμοδοτήσεις. Πρόταση ε, κανονισμού του Συμβουλίου για συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων φυσικών ή νομικών προσώπων, οργανισμών και φορέων ως προς την κατάσταση στη Σομαλία. Ε, θα κάνουμε γνωμοδότηση για το ίδιο θέμα ε, σχετικά με τη Συμπάμπουε για να μπορέσουν να παγώσουν ορισμένα στοιχεία ενεργητικού και ε, να απαγορευτεί η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων προσώπων. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνουμε γνωμοδότηση εμείς. πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για να τροποποιεί τον κανονισμό σε σχέση με την ίδρυση χρηματοπιστωτικού μέσου για τη συνεργασία με τις βιομηχανικές χώρες και άλλες χώρες υψηλού εισοδήματος ICI και, και, και κάποια άλλα εδάφη. Πρόταση κανονισμού ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού ε, σχετικά με την ίδρυση ε, σταθεροποιητικού μέσου. Την έκθεση αυτή θα την καταρτήσει η πρόεδρος και πάλι χωρίς ε, καταβάλει κανένα πόντο. Ομάδες εργασίας τώρα. Κάθε ομάδα εργασίας θα έχει έξι πλήρη μέλη και έξι αναπληρωματικά. Ε, η ε, Επιτροπή Εξωτερικών και Αντιπροσωπείες καλούνται να στείλουν μέλους τους σε κάθε συνεδρίαση της ομάδας εργασίας με καθεστώς συμβουλευτικό. Οι πρόεδροι έχουν οριστεί ε, με το σύστημα ε, σοσιαλιστές ε, ΕΛΚ, σοσιαλιστές ε, D και ΕΛΚ για τις έξι ομάδες και ο αντιπρόεδρος θα είναι κάθε φορά από άλλη πολιτική ομάδα, διαφορετική του προέδρου και κατά προτίμηση από μικρότερη ομάδα. Ο κύριος Δίβα. Πρόεδρε, μπορώ να διορθώσω κάτι, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε για το μέσο, ε, όχι το DCI για την οικονομική συνεργασία, θα γίνει από τη δική μου ομάδα και δώσαμε και πόντο για να πάρουμε την έκθεση αυτή. Yes, it was... yes, you're right. Έχετε δίκιο. Uh, okay. Uh, ECR uh, e είναι η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Το σημειώνουμε και λαμβάνετε υπόψη ε, στο έγγραφο. Θα το διορθώσουμε. Σας ευχαριστώ. Ε, ήμουνα στους αντιπροέδρους. Η εντολή είναι για δυόμιση χρόνια των ομάδων εργασία και κάθε ομάδα εργασία εγκρίνει και υιοθετεί τη μέθοδο εργασίας του. Θα έχουμε μόνιμο εισηγητή για την ανθρωπιστική βοήθεια. Εγκρίθηκε ένα σχέδιο εντολής. Η ομάδα εργασίας για τον προπολογισμό θα είναι ανοιχτή για όποιον ενδιαφέρεται όποιο μέλος της Επιτροπής μας θέλει να, παρακολουθεί τις εργασίες για τη Συμφωνία Κότονου και τις διαπραγματεύσεις, θα υπάρχει τακτική ε, συνεδρίαση ε, από τώρα μέχρι το Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων μας για ανταλλαγή ε, απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Για το 2009 τώρα αποστολές, δύο μέλη στο Μπαγκλαντές για να μελετηθεί ο τρόπος ε, με τον οποίο λειτουργεί το DCI και η διευκόλυνση επιστημιστική σε μια χώρα που ε, πλήττεται σημαντικά από τις κλιματικές αλλαγές. Το κυλιόμενο σύστημα DONT χρησιμοποιείται και πάλι για τη θέση αυτή. Ένας θα είναι από το ΕΛΚ και ένας από τους πρασίνους ε, στην αποστολή αυτή. Και τώρα αποστολή παρακολούθησης του GPI ε, δύο φορές από πέντε μέλη. Πρώτη προτεραιότητα και αποστολή είναι η Ζιμπάμπουη και δεύτερη η Μποτσουάνα. Και η Ναμίμπια ενδεχομένω. Το κυριαρχημένο σύστημα DONT επίση χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθεση των επιτροπών αυτών. Ένας από το ΕΛΚ, δύο σοσιαλιστέ, δύο ΑΛΔΕ και ε, ένας από το ECR για τη Ζιμπάμπουε, Ποτσουάνα, ένας ΕΛΚ, τρεις σοσιαλιστές, ένας πράσινος. Όλα τα μέλη θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει και ε, στην αντίστοιχη δικασία για την Αγγόλα. Τώρα, ποσοστώσεις για τις αποστολές θα προσπαθήσουμε να ε, εγκριθεί η ποσόστοση που δεν έχει καλυφθεί από την προηγούμενη ε, θητεία για να στείλουμε και τρίτο μέλος στο Μπαγκλαντές. Και αν εγκριθεί αυτή η θέση θα την πάρουν φιλελεύθερη. Προσπαθούμε να πάρουμε έγκριση και άδεια επίσης για να χρησιμοποιήσουμε ε, και την ποσόστοση της παλιάς Επιτροπής για να στείλουμε ένα μέλος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σε κοινή αντιπροσωπεία με ε, την Επιτροπή Εξωτερικών τον Οκτώβριο και ε, θα ε, στείλουμε και αποστολή παρατήρησης εκλογών στη Μοζαμβίκη. Οι βουλευτικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου και κανονικά θα πρέπει να είναι ε, προτεραιότητα για αποστολή παρατηρητών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά ορίσαμε και τις ακροάσεις για το υπόλοιπο του έτους. Πλήρες ακροάσεις μπορούν να γίνουν μόνο στις τακτικές μας συνεδριάσεις ε, σε δύο μισές μέρες, 9 και 10 Νοεμβρίου. Αντίκτυπος παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, με εμπειρογνώμονες είναι η ακρόαση αυτή. Οι εμπειρογνώμονες που θα προσκληθούν είναι ο Τζέφρι Σάξ, καθηγητής από ε, το London School of Economics και οι ομάδες θα προτείνουν άλλους δύο εμπειρογνώμονες γραπτός. Οι ομάδες επίσης μπορείτε να κάνετε τις προτάσεις σας για τις ακρόασεις του 2010 μέχρι την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών με ε, θέματα και εμπειρογνώμονες ε, ε, για σύντομες ε, συνεδριάσεις και συζητήσεις ενδεχομένως και εμπειρογνώμονες με αντικρώμενες απόψεις. Και συνεργασία επίσης με το ελεκτικό συνέδριο κοινή ακρόαση ή ακρόαση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Έχουμε δύο μελέτες ε, που έχει αναθέσει η προηγούμενη Επιτροπή το 2009 για την υποστήριξη ε, μακροοικονομική και την αποναρκοθέτηση της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτά θα τα συζητήσουν ξανά οι ε, συντονιστές στις 5 Οκτωβρίου. Επίσης, θα κάνουμε κοινή ακρόαση με την κυρία Σαΐτ μαζί με την Επιτροπή ε, Εξωτερικών στις 10 Σεπτεμβρίου. Εκπροσώπηση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κέντρο Βορρά Νότου θα είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα. Αν έχουμε περισσότερες υποψηφιότητε από τις θέσεις, θα το συζητήσουν και θα ψηφίσουν οι συντονιστές στην επόμενη συνεδρίαση για να επιλέξουν δύο πλήρη μέλη μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών και το Γραφείο των Βρυξελών στις 28 Σεπτεμβρίου θα παρετεθεί κοινή δεξίωση. Κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών θα έχουμε στις 12 ε, Οκτωβρίου με τον κύριο Ροσμισήρο, ε, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Έχουμε εξαμηνιές ε, συνεδριάσεις ε, για τους συντονιστές, για το προσωπικό, για τα μέλη. Επίσης θα πρέπει να ορίσουμε αντιπρόεδρο με ειδική αρμοδιότητα για το gender mainstreaming, η κυρία Κρέτσου, για δυόμιση χρόνια και πρωτοβουλία για προφορική ερώτηση και ψήφισμα για ε, τη διάσκεψη της Κοπενχάγης στο ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Προφορική ερώτηση και σχέδιο ψηφίσματος όπως έχει σχεδιαστεί. Διατηρείται το αίτημα για εξαχωριστή συζήτηση στην Ολομέλεια για τις συνέπειες ε, της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Νομική γνωμοδότηση για τη συμφωνία την αλευτική με το Μαρόκο κλεισμένων των θύρων, ανταλλαγή απόψεων με ε, τη νομική υπηρεσία για να αποφασιστούν ενδεχόμενα νέα μέτρα μετά την ανταλλαγή απόψεων. Ανταλλαγή απόψεων με τη Μαυριτανία, με εκπροσώπους του Συμβουλίου και για τις εκλογές στο Αφγανιστάν, ιδιαίτερα ε, η επίπτωσή τους στην αναπτυξιακή συνεργασία. Κατά προτίμηση κοινή συνεδρίαση ε, με την Επιτροπή Εξωτερικών. Η Επιτροπή μας θα ζητήσει ε, η αποστολή αντιπροσωπεία για το Κάρδιβ να είναι 14 μέλη, 14, ε, τα μισά από την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου και τα μισά από την Επιτροπή μας που συμμετέχουν στην κοινή συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Θα δούμε ποιο θα είναι το μέγεθος ε, της ε, αντιπροσωπείας, θα το αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων. Εκτός και αν ε, συμφωνήσουμε εμείς με την Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου και το δεχτούν οι συντονιστές. 18 σημεία ήταν μακροσκελέστατη αυτή η αναφορά. Έχετε ζητήσει το λόγο. Πρόεδρε, δεν θέλω να καθυστερήσουμε περισσότερο τη συζήτηση. Δεν θέλω να το να ανοίξω το θέμα, αλλά απλώς ήθελα να πω ότι ε, σύμφωνα με τον κανονισμό υπάρχει ένας συντονιστής ανά ομάδα και αν ακολουθήσουμε τον κανονισμό θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, συντονιστής. Αυτό θα το πούμε και στη διάσκεψη των Προέδρων η ομάδα μου γιατί δεν συμφωνούμε καταρχάς με αυτή την πρακτική. Αλλά ούτως ή άλλως εφόσον το ζητήσετε στη συνάντηση των συντονιστών θα το συζητήσουμε τώρα. Οι κανονισμοί δεν λένε κάτι τέτοιο λέει ο κύριος Μίτσελ. Λέει may have, μπορεί να έχουν. Το συζητήσαμε και στην ομάδα μας εάν οι σοσιαλιστές θέλουν να προχωρήσουν από εδώ και πέρα έτσι ε, μπορούν να το κάνουν αλλά επειδή και εγώ έχω θητεύσει σε αυτή την επιτροπή ε, προσπαθώ να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός Είμαστε μεγαλύτερη ομάδα από εσά, επομένω ε, θα πρέπει να, να λάβετε κι εσεί τι ευθύνε σα και τι συνέπειε. Λοιπόν, δεν θέλουμε να ακούμε όλα αυτά τα μεγάλα λόγια, ε, γιατί στο κάτω-κάτω και αυτοί που τα λένε θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να δεχτούν τι συνέπειε των όσων λένε. Κοιτάξτε, είχαμε συζήτηση των ε, συντονιστών, λέει η Πρόεδρος. Κοιτάξτε, πρέπει να σταματήσουμε. Έχουμε, ε, ε, είναι πολύ βεβαρημένη η μερίσια διάταξη και πρέπει να προχωρήσουμε. Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι περιτό να ξεκινήσουμε τώρα να προσβάλλουμε ο ένας τον άλλον. Δεν είναι επαγγελματικό αυτό. Κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μίτσελ, κοιτάξτε, κοιτάξτε, μέχρι τώρα Ακούσαμε για τη Ρωμα, Εκκλησία, για το Βατικανό. Για Λοιπόν, εδώ μιλάμε, ε, εκφράζουμε τις απόψεις μας και δεν χρειάζεται να γίνονται τέτοια σχόλια επιπροσωπικού χαρακτήρα. Πολύ ενέργεια, λέει η πρόεδρο, σε αυτή την αίθουσα. Μήπω θα μπορούσαμε την ενέργεια αυτή να την διοχετεύσουμε σε πιο ε, θετικά κανάλια, τέλο πάντων, με πιο θετικό τρόπο να την χρησιμοποιήσουμε. Τέλος πάντων, ελπίζω ότι όλοι έχετε την κάρτα για τις ψηφοφορίες. Ξέρετε πως, θυμόσαστε πως πρέπει να ψηφίσουμε. Πρέπει να κάνει κλικ η κάρτα μπαίνοντα στο μηχάνημα. Έχετε τρία κουμπάκια. Με το πρώτο ψηφί, υπέρ ψηφίζετε, το δεύτερο αποχή και το κόκκινο είναι ε, ψηφίζετε κατά. Θα κάνουμε μια δοκιμή. Να κάνουμε μια δοκιμή. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Βάλτε την κάρτα σας. Και μετά δοκιμάστε τα, τα κουμπάκια. Yes, in the middle. Okay, the boot is closed. Okay. We are doing a secret vote here. Είναι ε, μυστική ψηφοφορία εδώ. Ναι, ναι, μυστική ψηφοφορία. Okay, now we We have it. it try again. Λοιπόν, ας το ξανακάνουμε. Ας ξαναδοκιμάσουμε. No, ça marche pas. Non, ça, vous l'avez fermé, là, avec ça. Pour, pour l'ouvrir, c'était ça. Voilà, ça, c'est Donc, on Maintenant, on can vote. We vote. Now it's open. This is... Now it's working. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα λειτουργεί. Σωστά. Και μετά φαίνονται και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην, στην οθόνη.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 will be registered. won't appear in any. Yes. Okay. Then we will start. Λοιπόν, ξεκινάμε. Και ψηφίζουμε πρώτα απ' όλα τις τροπολογίες στην προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Όπως τροποποιείται από πολλά μέλη της Επιτροπής μας. Αλλά αναγράφεται μόνο το όνομα του κυρίου Πεγιών στην τροπολογία αυτή. Πρέπει να σας πω ότι την έχουν συνυπογράψει πολλοί. Και εγώ προσωπικά, η κυρία Λιωτά, η κυρία Ντεσαρνές, ο κύριος Κονβεντίτ, ο κύριος Μπένα η κυρία Τροτμάν, ο κύριος Μπέρμαν, ο κύριος Σασόλη, ο κύριος Μαρτίνεθ, ε, η κυρία Ντεκεζέρο, ο κύριος Τριολιά, ο κύριος Κάσμαν, ο κύριος Δερόσα, η κυρία Σαργεντίνη, η κυρία Τόγια, η κυρία Γκρέσ, ο κύριος Δεζίρ, ο κύριος Στάς και ο κύριος Αρίφ. For... Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία αυτή. Okay. And it's closed. They, are, they have problems. Problem? What's the problem? Yes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 yes. Okay. Λοιπόν, τι προβλήματα έχετε. Έχετε πρόβλημα. Oh shit. Υπήρξε πρόβλημα με ένα μηχάνημα και μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Ήταν η πρώτη. Λοιπόν, άρχεται τώρα η ψηφοφορία για την πρώτη τροπολογία στην προφορική ερώτηση. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. πέρα στι ψηφοφορίε. Εγκρίνεται λοιπόν. Τώρα θα ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αντίστοιχες τροπολογίες. Έχουμε την τροπολογία υπαριθμών 1. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Μια στιγμή. Δεν ξέρω, σηκώνετε χέρια. Ε, τι θέλετε να πείτε, ζητάτε το λόγο, λέτε ότι δεν δουλεύει το μηχάνημά σας. Όχι. Καμιά φορά ε, υπάρχει ένα μέλος που σηκώνει το αντίχειρά του για να δείξει στους άλλους τι θα ψηφίσουν υπέρ ή κατά. Γουίπ. Α, αρχάρια είμαι. Κάθε φορά που έβλεπα χέρια νόμιζα ότι έχετε πρόβλημα ζητάτε το λόγο. Όχι, όχι, δίνουμε γραμμή στα μέλη μα. Ωραία. Σα ευχαριστώ πολύ που με ενημερώνετε. Πέρα. So Εγκρίθηκε. Επόμενη ψηφοφορία τώρα. τροπολογία του κύριου Πεϊό. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε για το ψήφισμα. Πολλές τροπολογίες. Α, συγγνώμη, μου λέει η γραμματεία ότι πρέπει να ψηφίσουμε το τελικό κείμενο της προφορικής ερώτησης όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει λοιπόν τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Τι ψηφίζουμε, λέει ο κύριο Μίτσελ. Ναι, έχει επικρατήσει μια μικρή σύγχυση. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα το τελικό κείμενο τη προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπω τροποποιήθηκε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στο ψήφισμα. Ο κύριος Μπέρμαν. 29 με 34 παρακαλώ μπορούμε να ψηφίσουμε. Έχω και μια προφορική τροπολογία λένε οι πράσινοι.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 Τι είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Α, εγκρίνεται ομόφων. Η τροπολογία υπαριθμό 30. Ζολή και Λέριξ Αρζεντίνη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Η 31 μια προφορική τροπολογία έχουν εδώ οι πράσινοι. Ναι, θα θέλαμε να αλλάξουμε must be integrated to να γίνει must not be dissociated from στα αγγλικά. Αυτή η προφορική τροπολογία. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Πέρας. Πολύ γρήγορα πάμε. Όχι, εντάξει. 20. Να εγκρίνεται μου Η τροπολογία υπαριθμών 32. Σας ρώτησα αν μπορούμε 32, 33, 34 να τις ψηφίσουμε μαζί, λέει ο κύριος Μπέρμαν. Σας ευχαριστώ για την πρότασή σας. Πολύ καλή ιδέα. Ψηφίζουμε λοιπόν την 32. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Αγκρίνεται. 33 υπέρ. Όχι, αρχίζει η ψηφοφορία, συγγνώμη. Ψήφισατε όλοι. Πέρασα. Εγκρίνεται. Η 34 αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Συγγνώμη, έγινε ένα λάθος. Όχι ακόμα. Ψηφίσατε όλοι. Δεν έχει αρχίσει ακόμα. Τώρα αρχίζει. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Η 35 Το κύριου Αρσένη with much. Μάλιστα. Πρέπει να την ψηφίσουμε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Everybody has voted. Vote is closed. Αν ψηφίσατε όλοι πέρας. Η τροπολογία 36, Ρινάλντι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Everybody Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 37, Γκέρενς. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα. Εγκρίνεται. Η επόμενη τροπολογία υπαριθμό 38 καταπίπτει, διότι εγκρίθηκε 32. 39. Τυρολιάντε Σιρ γιόν 39. Ψηφίζουμε παρακαλώ αρχής ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 40. Κασμαρέκ. Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα. Εγκρίνεται, λέει η πρόεδρο. Ενώ έχει απορριφθεί. Δηλαδή απορρίπτεται. Η 41 έχει αποσυρθεί. Η 42 του κυρίου Πεγιό πρέπει να ψηφιστεί. Αρχίζει ψηφοφορία για τη 42 του κυρίου Πεγιό. Ψηφίσατε όλοι ή πέρασε. Εγκρίνεται. 43. Λέει εδώ ότι καταπίπτει αν εγκριθεί 40 ή 41. Άρα καταπίπτει. Όχι. Πρέπει να τη ψηφίσουμε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Είναι 44. Ζολή και Λέρκες Σαρζεντίνη, αρχή ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 45 της κυρία Στόγια. Αρχή υποφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 46. Ζολί Κέλλερ και Σαρτζεντίνη. αρχη πληροφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 47. Τυρολιάντε Ζερπεγιόν. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία υπαριθμών 48, Κασμαρέκ. Άρχισε ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 49. Αρχή ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η 50 της κυρίας Τσίμα αρχή τώρα ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Amendment 51. 51. Έρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Πενήντα δύο. Αρσένη. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η επόμενη αποσύρεται 54 της σήμερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. 55 Τζόλι Κέλλερ Αργεντίνη, άρχιτε ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Στην 56 έχει ζητήσει η κυρία Σαρκεντίνη σε τμήματα ψηφοφορία. Και έτσι πρώτα θα ψηφίσετε, πρέπει να το διαβάσω. Όχι, έχετε το κείμενο. Το πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. δεύτερο, ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Okay. 57 δεκάισερ, άρχεται η ψηφοφορία. Άχι ψηφοφορία. Ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. 58. Δεκάιζερ. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 59. Κάσμαρεκ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. Yes, now we got to the recitals and citations. Uh, amendment 3. Στην επόμενη, συνεδρι... Στην επόμενη τροπολογία υπερθυμών 3 Αρσένη, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 4 τροπολογία. Ζολή Κέλλερ Σαρκεντίνη, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι υπέρ ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 5. Τζόλι και στην Αργεντίνη, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρα στις ψηφοφορία. Εγκρίνεται. μόνο έξι Ντέβα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ο φορέας. Εγκρίνεται. Επτά. Του κύριου Τίβα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε. Να τα δούμε αν μπλοκ όλα. Α, έχει αποσυρθεί η επόμενη. 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Δέκα. Γιατί η 9 έχει αποσυρθεί. Στη 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Στην 9. Ψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται. 11. Ντέβα. η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται. Η ψηφοφορία λέει η πρόεδρος. Α, κλείνει η ψηφοφορία και απορρίπτεται. Μπορούμε να ψηφίσουμε on αν θέλετε. 12, 13, 14. Όχι, δεν θέλετε. 12 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Και ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Adopted. Amendment Εγκρίνεται. Στη 13, Δεκάιζερ, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της προφορίας. Εγκρίνεται. 14. Δεκεζέχ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 15 Δεκεζέχ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 16. Ζουλή Κέλλερ Αργεντίνη, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεν. Άρχιτη ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 18. Δέβα. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 19. χωριστά την κάθε τροπολογία. 19, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήψαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 20, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 με 24 μπλοκ, συμφωνούν όλοι. Πολύ καλά. 21 24 μαζί. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνονται. 25. Σόλιο και Λέξα Αργεντίνη. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τη Βολέντα Ζήρπελιό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27 των ιδίων άρχεται η ψηφοφορία. 27 όπως είπαμε. Εψήφισαν όλοι πέρα της Εγκρίνεται. 28 έχει αποσυρθεί. αριθμό 1 Τσίμερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δύο ντεύω Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. So, I, yes, by last a little bit. Okay, so uh, vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία στο τελικό κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το κείμενο. Λοιπόν, τώρα θα ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση. Δεν θα ήταν πιο σύντομα ψηφίζουμε με διανατάσεις χειρός και αν υπάρχει καμία ε, αμφιβολία να κάνουμε ηλεκτρονική. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες ακόμα. Συμφωνώ, λέει ο κύριος Μίτσελ. Θα ήταν πιο γρήγορο. Είναι πιο γρήγορο. Και πρέπει να φύγουν και οι διερμηνείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος, για το εξαιρετικό τους ε, έργο, οι οποίοι όμως σχολάνε αυτή τη στιγμή και θα φύγουν και θα συνεχίσουμε χωρίς διερμηνία